Mes chers collègues, nous voici αυτή την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ε, Προπολογισμών και Ελέγχου Προπολογισμού. Για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρόκειται για την ε, απλούστευση του δημοσιονομικού κανονισμού. Κοινή επομένω ε, συνεδρίαση και σκοπό μας είναι να συνεχιστεί η εξέταση της ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Νοεμβρίου και αφορά τον δημοσιονομικό οργανισμό ο οποίο ε, πρόκειται να ισχύσει για τον ε, προπολισμό της Αυτό θα γίνει σε δύο μήνες. Πρώτα πρώτα θα έχουμε παρουσίαση του σχεδίου κειμένου της εκθέσεως από τους δύο συνεισηγητάς, την Ίγκε Γκρέσλε και τον Ρίτσαρντ Ashworth. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανταλλαγή απόψεων παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ελληνικού Συνεδρίου. Στη συνέχεια δε, από τις 3 ώρα δηλαδή, πρόκειται να έχουμε ένα εργαστήρι και θα ακούσουμε τη γνώμη του, του Ελληνικού Συνεδρίου, γενικέ παρατηρήσει, αλλά επίση και διάφορου ομιλητέ που έρχονται από πολλέ διαχειριστικέ αρχέ, φορεί, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει για συγκεκριμένα ζητήματα. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω από πλευρές διαδικαστικής ότι η έγκριση του οριστικού κειμένου προβλέπεται για τις 11 Πέμπτου. Επομένως, έχει καθοριστεί προθεσμία για τις ε, τροπολογίες και είναι η 6η Απριλίου το μεσημέρι. Ήδη οι συνεργαμόδιε επιτροπέ έχουν εξετάσει μια πρώτη εκδοχή του κειμένου και πρόκειται ε, προσεχώ να γνωμοδοτήσουν οριστικά και έχουμε πέντε τον ρόλο τη ε, συναρμοδίας επιτροπή δυνάμει του άρθρου 54 με συγκεκριμένε αρμοδιότητες ενισχυμένε βάσει του πρωτοκόλου όπω αυτό επικυρώθηκε από τους Προέδρους ε, Ρέτζι, Εμπλουά, Τραν και Ήτρε. Επίσης σα υπενθυμίζω ότι οι σκιώδες ηγητέ από τι πολιτικέ ομάδες για τις Επιτροπές Προπολογισμών και Ελέγχου είναι για τους σοσιαλιστές ο Βλαντιμίρ Μάγκα και η Νιέσα Γιάλα Σέντερ. Για το Λαϊκό Κόμμα ο κύριος Σαρβαμά, για τους ε, ελευθέρους ο Νάσμπι Αλή, για τους ε, πράσινου, ο κύριος Τάραν και ο κύριος Στάς, για την Ενωτική Αριστερά και για το EFDD ο Μάρκο βάλει. Αρχίζουμε. Αν δεν έχει την αντίρρηση, να ακούσουμε τους δύο συνεισηγητάς. Κυρία Πρόεδρε, συνεισηγήτρια, αρχίστε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να καλωσορίσω τα μέλη της Επιτροπής Έλεγχου του Προπολογισμού επίσης. Είμαι της Επιτροπής Έλεγχου του Προπολογισμού ασχολούμαστε με αυτό το θέμα εδώ και καιρό. Θέλω να ευχαριστήσω τους Κιώδης και να πω ότι πρέπει να έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ επιμελείς και συνεχίζεται ε, είναι απαραίτητο να είμαστε ακόμα περισσότερο επιμελείς. Πρέπει να δούμε αυτήν την ε, αξιολόγηση γιατί άλλαξαν όλα αυτά τα πράγματα εγώ χρειάστηκε να αναζητήσω τα παλαιά κείμενα, τα παλαιά τμήματα και να δω τι περιλαμβάνεται και τι δεν περιλαμβάνεται στο νέο κείμενο και αν δεν περιλαμβάνονται κάποια τμήματα γιατί δεν περιλαμβάνονται. Έχουμε ε, το detection. το πάνελ οικονομικών παρατυπιών Είχαμε και το ελεγκτικό συνέδριο που είπατε αυτό το πάνελ ε, έχει διάφορες αρμοδιότητες. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρμοδιότητα της κάθε αρχής και γι' αυτό αναδρομικά καταστήσαμε σε ισχύ αυτό το τμήμα. Έχουμε τραπε... πολλές τροπολογίες, ορισμοί, νέοι ορισμοί για τα commitments, για τις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων και την υλοποίησή τους. Εμείς προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε όλες τις αμοιότητες ε, που μας δίνει ο κανονισμός ε, για την Επιτροπή μας. Έχουμε κάποιες αρμοδιότητες που παλιά είχε η Επιτροπή Προϋπολογισμών μετά την Επιτροπή με τη συζήτηση με τους Κιώδης αποφασίσαμε όμως να ξαναδώσουμε αυτές τις αρμοδιότητες στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Δεν νομίζω ότι εμείς ε, βέβαια μπορούμε να απο... απεμπολούμε κάποια δικαιώματα. Ξέρουμε ότι μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά οι συνάδελφοι αυτά τα δικαιώματα. Πάντως υπάρχουν τα δικαιώματα και δεν πρέπει να τα απεμπολούμε. Γιατί αυτό μας διευκολύνει και τη ζωή των να υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα. Και δείχνουν όλα αυτά πόσο δύσκολη είναι όλη αυτή η διαδικασία. Ιδίως ό,τι αφορά την απλούστευση δεν δεχτήκαμε λοιπόν την αλλαγή ε, και για διάφορες άλλες διατάξεις ε, δεν τις ε, κάναμε δεχτές. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις οι οποίες έχουν εξαφανιστεί, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Γιατί υπάρχουν σημαντικές οδηγίες πολύ ακριβή για τη διαχείριση των προγραμμάτων. Οι διαχειριστές των προγραμμάτων πρέπει να έχουν αυτές τις οδηγίε. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν εξαφανιστεί λοιπόν οι διατάξει που αφορούν ε, τι οδηγίε προς τους διαχειριστές των προγραμμάτων. Προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο δυνατόν πιο ξεκάθαρο το κείμενο της Κομισιόν και φαντάζομαι ότι θα βοηθήσουν και οι συνάδελφοι προς αυτό το σκοπό σε ό,τι αφορά την αναφορά, το reporting, τα χρηματοδοτικά μέσα. Έχουμε ε, κάνει τα θέσεις τροπολογίες για τα service level agreements, ότι θα μπορούσαν γενικέ διευθύνσει να αποφασίζουν, να, να παίρνουν αποφάσεις, να αφαιρούν κάποιες, ε, κάποια κάποια τμήματα και αυτό προσπαθήσαμε να το αποτρέψουμε. Έχουμε κάνει επίσης κάποιες άλλες ε, προτάσεις για νέες μορφές χρηματοδότησης ε, και για τις εταιρικές σχέσεις. Ε, θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ως προσανατολισμός στις επιδόσεις, καλύτερη αξιολόγηση η Αντιπρόεδρος Γεωργίευα μας είχε πει ότι και ένα αναθεώρηση του κανονισμού θέλει να ενισχύσει το σκέλος των επιδόσεων. Αναφερόταν σε μια-δυο παραγράφους το θέμα, αλλά όχι πάρα πολύ αναλυτικά, γι' αυτό προσπαθήσαμε να ε, το κάνουμε εμείς ακόμα πιο ξεκάθαρο. Μετά από μακρές συζητήσεις που είχαμε με τους σκιώδες, ό,τι αφορά τα καταπιστευματικά ταμεία, που θέλει η Επιτροπή να επιτρέψει να δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχει αυτός ο περιορισμός εντός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εμείς θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος ε, από τη δική μας πλευρά. Δηλαδή, θέλουμε να δίνουμε τη σύμφωνη γνώμη μας, να υπάρχει διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι αυτά τα καταπιστευματικά ταμεία ανήκουν στου δορυφορικού αυσεκτελεστικού οργανισμού και εμεί δεν έχουμε κάποιο δικαίωμα. Έχουμε πάρει επίση κάποιε συστάσει ε, υπόψη μα από το ελεγκτικό συνέδριο, το δεύτερο τμήμα ε, της έκθεσης ε, και σε ό,τι αφορά τις επιτροπέ του εσωτερικού ελέγχου. Μιλάμε για, υποστηρίζουμε τον ενιαίο έλεγχο, τον ενιαίο λογιστικό έλεγχο, single audit, μελετάμε τις διάφορες μεθόδους χρηματοδότησης. Αν έχουμε 50% επιδοτής 10% χρηματοδοτικά μέσα, θέλουμε να ισχύσει το πρώτο και το δεύτερο. Και νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση. Γνωρίζω ότι μπορεί να μην έχετε εξοικειωθεί απόλυτα με αυτές τις τροπολογίες. Έχουμε όμως και το τριμερείς διαλόγους. Και πρέπει να πω ότι και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν ήταν τόσο, δεν μας ήταν τόσο οικία. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τη διαχείριση, θέλουμε να είναι διαχείριση των κονδυλίων άμεση και σε ό,τι αφορά την ανακατανομή. Θέλουμε να συναποφασίζει Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. και δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον να ανακατενέμονται πόροι και να πηγαίνουν από άλλα ε, κονδύλια, από άλλα πράγματα στο ΕΦΣΥ. Έχουμε και τον κανονισμό για τα διευρωτικά ταμεία. Είναι το δεύτερο τμήμα αυτό αυτής της διαδικασίας. Για το cross-reliance verification στηρίζουμε αυτές τις ε, αρχές αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε την επαλήθευση των διαφόρων εταίρων σε ό,τι αφορά δε την υποχρέωση αναφορών ε, υποβολής εκθέσεων από την Κομισιόν. Θα πρέπει να ξέρουμε τις πληροφορίες που θα πρέπει εμείς ε, να λαμβάνουμε Υπάρχει μια πρόταση που αναφέρεται στην έκθεση, αλλά δεν νομίζω ότι ρυθμίζει όλα τα προβλήματα και καθαριστά ξεκάθαρη αυτή την υποχρέωση της Κομισιόν για υποβολή εκθέσεων. Επίσης για απαγόρευση των ε, ιονί των εικονικών εταιριών. Χαιρόμαστε για την ε, πρόταση και καλό θα ήταν να υπάρχει ε, συγκεκριμένη αυτή διάταξη. με το non-profit, τη μία αποκόμιση κέρδους δηλαδή, είναι μια αρχή την οποία έχουμε συμπεριλάβει. Η αρχή λοιπόν της μία αποκόμισης κέρδους θέλουμε να καταργηθεί, συγγνώμη. Είδαμε κάποιες κοινωνικές μικιώσεις σήμερα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση. Και νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει ο κλάδος αυτός και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα κάνει κάθε προσπάθεια. Θέλω να βοηθήσω και τον συνάδελφο Άσχουερθ. Είναι πάρα πολύ ευρύς ο φάκελος. Θα ιδρώσουμε, πιστεύω, απέναντι στο Συμβούλιο. Ελπίζω να περάσουν οι δικές μας ε, τροπολογίες. Και ελπίζουμε επιτακές και στο πλαίσιο των δημερών διαλόγων να έχουμε ένα καλό ε, αποτέλεσμα. Υπάρχουν πράγματα που θα ήθελα να είναι διαφορετικά. Δηλαδή να υπάρχουν τροπολογίες που θα προωθούν ακριβώς αυτό το στόχο της απλούστευσης και όχι να αλλάζουν όλα αυτά. Να έχουμε δηλαδή όλη αυτή, όλες αυτές τις αλλαγές. Έχω επενδύσει πάρα πολύ, έχουμε επενδύσει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι άξιζε, το λέω ξεκάθαρα, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη από την πρόταση Κομισιόν. Ε, αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον συνεισηγητή μου. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Γκλέσσερ και για την πραγματογνήμησή σα και να σα πω πω κατά κάποιο τρόπο είστε η συλλογική μνήμη αυτού του κανονισμού και νομίζω πως τα δικά σα λόγια ουσιαστικά μας οθούν στο να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δείξει τα δικά της χαρτιά. Τώρα δεν ξέρω τι πιστεύει όλο αυτό ο κύριος Ashworth. Έχετε το λόγο πάντως, συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τη συνεισηγήτριά μου όχι μόνο γιατί είπα όσα θα έπρεπε να έχω πει εγώ, οπότε με διευκολύνει πάρα πολύ στο έργο μου, αλλά και γενικότερα. Να σας πω ότι καταρχήν εμείς καλωσορίζουμε αυτή την κατεύθυνση που ακολουθεί στις περισσότερες από τις προτάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω, όπως είπε και η συνάδελφος, πως αν ε, στόχος αυτός ήταν να μειωθεί ε, και το ποσοστό σφάλματος και το διοικητικό βάρος και ε, να μας δώσει περισσότερα και πιο απτά αποτελέσματα και σε επίπεδο παραδοτέων στους δικαιούχους, τότε ναι. Υπάρχουν όμως 4-5 σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Επιπτωσιολογική μελέτη. Λυπάμαι που δεν είχε ε, αρκετή επιπτωσιολογική μελέτη ή αξιολόγηση συνεπειών η πρόταση. Νομίζω ότι αυτό έρχεται και σε αντίθεση με τη διαθεσμική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία, οπότε το έχουμε ξαναβάλει εμείς στο κείμενο εν μέρη. Η κυρία Κρέσλε πολύ σωστά είπε πως χρειαζόμαστε μία κουλτούρα αποδοτικότητας. Αυτό ήταν εμβληματικό στοιχείο της πρότασης του προηγούμενου, της προηγούμενης Επιτρόπου Προϋπολογισμού, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε όταν ψάχνει κανείς λεπτομέρειες, πως όντως υπάρχει μία σύγκρουση μεταξύ της απλούστευσης και της ε, προετοιμασίας προϋπολογισμού βάσει αποδοτικότητας. Γιατί από τη μία έχεις ε, περισσότερους δείκτες αποδοτικότητας, το οποίο όμως ουσιαστικά δεν απλουστεύει το νομοθετικό έργο, αντίθετα. Οπότε εδώ έχουμε αρκετές παρατηρήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, πως θα πρέπει όλα αυτά να εσωτερικοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτό νομίζω ότι καλό θα ήταν ε, ε, να μας το πούνε αυτό οι, οι λογιστές οι οποίοι θα έκαναν ελεγκτικό, ε, θα παρουσίαζαν έργο για αυτές τις προτάσεις, ώστε να ξέρουμε τι μπορεί να μετρηθεί με ποιον δείκτη. Τώρα, η αρχή η, της, του μη κέρδους, δεν θα θέλαμε η απλούστευση να μην υποσκάπτει κάποιες παλαιές αρχές του, της σύνταξης προπολογισμού. Το συζητήσαμε με συναδέλφους, με σκιώθεις και δεν είμαστε σίγουροι και δεν μας πείθουν οι προτάσεις που καταθέτει για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν επανεισάγει μια σειρά παρατηρήσεων και βεβαίως αυτά θα δώσουν τροφή για πάρα πολλές συζητήσεις. Επίσης, εσωτερική έλεγχη και οι σχετικές διαδικασίες. Εμείς έχουμε ζητήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχουμε εισακούσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα όσα μας είπε το ελεγκτικό συνέδριο. Τι σημαίνει ο εσωτερικό έλεγχο και ποιε είναι οι σχετικέ διαδικασίε. Χρειάζεται η ξεκάθαρη η, ρύθμιση για το ποιο συγκροτεί αυτέ τι ομάδε, πώ εκπροσωπούνται και ποιε διαδικασίε ακολουθούν για συγκεκριμένε δράσει. Και το τελευταίο, υποβολή εκθέσεων και αναφορές. Και πάλι εδώ έχουν γίνει πολλές συζητήσεις με το ελεγκτικό συνέδριο και πρέπει να σας πω πως αυτό για το οποίο ανησυχώ εδώ και χρόνια είναι πως θέλουμε ο λογιστικός έλεγχος να μην αποτελεί απλή δήλωση συμμόρφωσης. Δηλαδή θέλουμε κάτι το οποίο θα δώσει περισσότερες προφορίες, θα μας κατευθύνει περισσότερο, θα είναι μια αναφορά με περισσότερο στοιχεία που θα είναι προς όφελος των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προτείνουμε λοιπόν το Ελληνικό Συνεδρίο να παρουσιάζει μια ενιαία ε, έκθεση που θα κάνει το λογιστικό έλεγχο μιας ευρύτερης γκάμας δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε ποιες δράσεις πλήττονται από παρατυπίες και θέλουμε και μια αναφορά σχετική με το τι γίνεται με τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Θέλουμε λοιπόν μια ενιαία, ενοποιημένη έκθεση. Είναι ένα ε, έγγραφο το οποίο έχετε μπροστά σας ε, και το οποίο έχει πάρα πολύ πλέον λεπτομέρειες με πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα όπως είπε και η συνάδελφος. Θα θέλαμε να μην είχαμε τέτοιους χρονικούς περιορισμούς αλλά καταλαβαίνετε πως ε, κάναμε αυτό που μπορούσαμε με τους πόρους που έχουμε και αυτό σας παρουσιάζουμε σήμερα. Bien. Merci. και ευχαριστούμε κύριε Άσχολος. Μας εξήγησαν οι συνεισηγητές μας την ουσία της νομοθετησής τους όσον αφορά την πλούστευση και απλοποίηση ε, του δημοσιονομικού κανονισμού, οπότε τώρα θα δώσουμε τη σκητάλη στους σκιώδεις συζητητές. Ο κ. Σαρδαμά για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα ειλικρινής ευχαριστίες προς τους δύο συζητητές αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο τους, μια που είναι γνωστή η σημασία του προϋπολογισμού όσον αφορά τη διαμόρφωση του μέντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά για όλο αυτό το, ε, το οποίο. Αλλά τέλος πάντων, για να δούμε τώρα την ουσία. Βεβαίως και εμείς ευθυγραμμιζόμαστε, είμαστε το ίδιο και είμαστε με τους συνεισηγητές και έχω να σας πω τα εξής. Οι προτεραιότητες μας Όσον αφορά αυτήν την αξιολόγηση και αναθεώρηση είναι πρώτα-πρώτα η απλούστευση, όπως ακριβώς είπαν και οι δύο συνεισηγητές, οι δύο δε, θα πρέπει να απλουστευθεί η ζωή των αποδεκτών. Το πιο σημαντικό αυτό είναι. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε compliance στα Οπότε και να προσέξουμε την πολλαπλή συμμόρφωση που είναι πολύ σημαντικό ορόσημο για την πορεία μας αλλά για να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες όσον αφορά αυτού του είδους τον προϋπολογισμό που βασίζεται στην επίδοση και απόδοση είναι δύσκολη υπόθεση αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι εάν είμαστε όλοι σύμφωνοι για το ότι θέλουμε να έχουμε σαν μπούσουλα στον προπολογισμό την απόδοση, τις επιδόσεις τέλο πάντων, θα πρέπει να δούμε ξανά αυτό το οποίο είπε ο κύριος άσχολη. Δεν ξέρω αν είμαι υπεραισιόδοξος. Αλλά ε, αν θέλουμε εξαντλητικά να ε, αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και να προχωρήσουμε σε απλούστευση αλλά και προϋπολογισμό που βασίζεται στα αποτελέσματα, ε τότε θα πρέπει να μειώσουμε αυτού του είδους την ερεσιμότητα; που έχει σχέση με τις δαπάνες. Διότι εξίσου με προβληματίζει το ότι εάν ακολουθήσουμε αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Δημοσιονομικό Κανονισμό κάνουμε όλε αυτέ τι ε, απαλληφέ και διαγραφέ που προτείνει, τότε ίσω το τέλο δεν είναι απλούστερο, αλλά απλώ θα δημιουργηθούν άλλου είδου προβλήματα. Αν όμω και επικεντρώσουμε την προσοχή μα, ούτω ώστε αυτή την αιρεσιμότητα για τι δαπάνε την προσέξουμε και να βγάλουμε δύο κουταλιές από αυτή τη σούπα και τόπιν ε, προσθέσουμε άλλες δύο που θα αφορούν όμως ε, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τότε ε, αυτό νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Και τι να σας πω, και εγώ τη πάω το μυαλό μου για να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Επίσης, ταυτόχρονα, για να δούμε τα έξις. Αν πει το Ελληνικό Συνέδριο, αλλά μου πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω, έχουμε εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου. Ναι, ναι. Νεύουν από τα πίσω έδρα, να εκπρόσωποι. Ναι, ναι, έχουμε, λέει ο Πρόεδρο. Γιατί δεν έχουμε πουθενά ορισμό των αποτελεσμάτων των επιδόσεων. Το Ελληνικό Συνέδριο μπορεί να μας προτείνει κάποιο ορισμό. Άλλη ερώτηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υιοθετήσει μία προσέγγιση επί τη βάση των κινδύνων. Επομένως αυτό θα να πω και όπως σας είπα επίσης να προσθέσουμε μια ακόμη μεταβλητή στο γύμνο που να έχει σχέση με τα, ε, με τα αποτελέσματα της επιδόσης. Αυτή είναι η συνταγή. Δύσκολη, δύσκολη μαγειρική λέει ο πρόεδρος και τώρα ο κύριος Μάνκα θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συνεισήγητές. Γνωρίζουμε πόσο πολύπλοκο ήταν το εγχείρημα, ότι ήταν πάρα πολύ ε, κουραστικές οι ώρες που χρειάστηκε να περάσουν. Και ιδίως εφόσον ούτε τότε ούτε τώρα δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις ε, αυτής της πρότασης της Κομισιόν. Ούτε και τι επιπτώσεις θα έχουν βέβαια και προτάσεις των δύο δικών, δικών μας γνωρίζουμε. Αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη την όλη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, αναθεώρηση, πιστεύω ότι έχει μια διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρηση ότι τώρα έχουμε απλούστευση 15 νομοθετικών πράξεων μέσα σε ένα έγγραφο. Και δεν έχουμε χρόνο, ενώ χρειαζόμαστε τον τριπλάσιο χρόνο αν θέλαμε να δουλέψουμε σωστά και με σοβαρότητα. Δυστυχώς όμως ενίοτε αυτό συμβαίνει. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν αναβολές γιατί ο στόχος είναι να μην γίνουν σφάλματα. Και η Επιτροπή μας, η ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θέλουν να λάβουν υπόψη ε, και τους στόχους για μη μείωση των κονδύλων του ορίζοντα 2020, σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τι αντίκτυπο θα έχουν όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες επιτροπές οι οποίες ε, γνωμοδοτούν, και τα κτλ. Αυτό που περιμένουν από μας ε, οι χώρες είναι ουσιαστικά να έχουμε υπόψη κατά συμφέροντα των αποδεκτών, των δικαιούχων, οι οποίοι αυτό που περιμένουν είναι καλά αποτελέσματα. Γιατί αν είναι καλά τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερη και η εφαρμογή, η υλοποίηση. Και αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να επαναλάβω ε, αυτό που είπε η συνάδελφος ε, Γκρέσλε, ότι δεν θα πρέπει τα διαθωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής ε, να το συγχέουμε με το ΕΦΣΙ. Έχουμε πόσο μας τι είναι το ΕΦΣΙ 2, το δεύτερο ΕΦΣΙ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η μεταφορά πιστώσεων, αυτή η ανακατανομή. Και νομίζω ότι ο φόβος μας είναι να εστίασε να περιοριστεί στις πιο πλούσιες περιοχές Λέει η Κομισιόν ότι τα συντηρητικά ταμεία ε, κινητοποιούνται εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά δεν το βλέπουμε να συμβαίνει στην πράξη. Τι γίνεται με τις χώρες συνοχής, για τις οποίες προβλέπεται η κατανομή των κονδυλίων. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μεταφορά κονδυλίων από τις ε, πιο φτωχές, τις πιο πλούσιες χώρες μέσω αυτής της ανακατανομής. Χαίρομαι που υπάρχει και πρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου, διαβάσαμε την έκθεση και την προσπογράφουμε. Θα περιμένω να ακούσω και τι θα υποθεί στο πλαίσιο του εργαστηρίου που θα ακολουθήσει Σημάθηκαν κάποια προβλήματα, συμφωνούμε. Αυτό που θα με ενδιέφερε όμως κυρίως να ακούσω είναι και η άποψη της Κομισιόν και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Φυσικά και είναι σημαντική απλούστευση. Αν επιστρέψουμε όμως αυτό που είσαι μέχρι τώρα, δεν θα προκύψει καμία απλούστευση. Η κατάσταση είναι πολύ πλοκή δεν θα πρέπει να απεμπολίσουμε τα δικαιώματά μας. Αλλά το να τα ανακαλέσουμε, να τα αποσύρουμε όλα ε, και να γυρίσουμε προς τα πίσω, δεν ξέρω κατά πόσο ωφέλει. Πάντως περιμένω να ακούσω πολύ ενδιαφέρον την Κομισιόν και βέβαια και το ε, σεμινάριο, το workshop που ακολουθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία ε, Αγιάλα Σέντερ δεν έχει έρθει. Ο κύριος Νίτς Μιαλή επίσης λείπει, δεν τον βλέπω. Ο Ιγμάρ δεν είναι εδώ. Ο Μπάρτ Στάς επίσης λείπει. Η κυρία Ριάντα δεν είναι εδώ. Ωραία. Αυτό ήταν ο κατάλογος ε, των ε, σχεδόν. Ο κύριος Βαντερ Κάμπ, νομίζω, από την Επιτροπή Τραν Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, Έχω την τιμή να είμαι ο συγκριτής δυνάμει του άρθρου 54 για την Επιτροπή των ε, Μεταφορών. Οπότε και εμείς ε, υποβάλαμε αυτή την γνωμοδότηση για την ε, έκθεση των συναδέλφων. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσουμε την κυρία Γκρέσλε και τον κύριο Άσφορντ για τη δουλειά τους, η οποία πραγματικά έγινε με μεγάλη ευσυνειδησία και ελπίζω ότι τελικά θα βγουν και οι μεταφορές κερδισμένες. Τώρα θέλω να σχολιάσω κάτι για την τροπολογία 4 αλλά και την υπαριθμόν 5 τροπολογίες και δύο της κυρίας Γκρέσλε άτυπα τα έχουμε πει και όσον αφορά την υπαριθμόν 5 λέει κυρία Γκρέσλε και από ε, επενδυτέ αλλά και χρηματοοικονομικούς φορείς και θεσμικά όργανα. Αυτή η φράση που έχει η κυρία Γκρέσλε νομίζω ότι θα μπλοκάρει πόρους που θα προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει κάποιο είδου διαχείριση αυτών των ε, πόρων. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Να δούμε επομένω πώ θα γίνει αυτό του είδου η διαχείριση των ε, ιδιωτικών πόρων. Θα πρέπει να την κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση ε, του ιδιωτικού τομέα στην χρηματοδότηση. Οπότε νομίζω θα πρέπει η κυρία Γκρέσλε να δει κάπως να χτενίσει αυτό το κείμενο και να αλλάξει αυτή τη διατύπωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ καταρχήν τους εισηγητές. Γιατί αφενός η Επιτροπή Προϋπολογισμού ήδη γνώριζε πως η τεχνική ποιότητα αυτής της έκθεσης θα ήταν εξαιρετική. Ξέραμε ποιος κάνει την εισήγηση. Νομίζω λοιπόν πως ήδη ξεκινούσαμε από αυτή την καλή αφετηρία. Τώρα, μείωση της γραφειοκρατίας, απλούστευση, αυτή είναι η οδός την οποία θα έπρεπε όλοι να ακολουθήσουμε και να περιμένουμε παράλληλα να βρούμε έναν τρόπο να χρησιμοποιούμε πιο σωστά τα κονδύλια που έχουμε με διαφάνεια σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι αυτή είναι μια σκέψη η οποία πάντοτε είναι παρούσα. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για τα διαστατικά ταμεία και για το ΕΦΣΕ και για τη διάκριση που μας ζητάτε να κάνουμε, να σας πω πως εγώ ανησυχώ κάπως. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες σύνδεσης όπου τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν και έχουν δεσμευθεί να χρησιμοποιήσουν ε, κονδύλια των Ταμείων Συνοχής και των Διευθυντικών Ταμείων για να δημιουργήσουν χρηματοπιστωτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε το να εργαστούν έτσι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα για το ΕΦΣΥ ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικά ή να υποκαταστήσουν τα ταμεία συνοχής. Αντίθετα θα πρέπει να συνδεθούν με όλα τα υπόλοιπα εργαλεία χρηματοδότησης που έχουμε και θέλω να σα δώσω ένα παράδειγμα. Αν έχουμε μία επένδυση στην οποία μόνο το ένα τμήμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα διαφθορτικά ταμεία. Το υπόλοιπο ή ένα άλλο τμήμα θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσω αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων, για παράδειγμα, αυτό το ε, Ταμείο ε, Ανάπτυξης που είναι το γνωστό πακέτο Juncker. Εμείς το χρησιμοποίησαμε και όπως στην Πορτογαλία χρησιμοποιούμε και τα Ταμεία Συνοχής. Γιατί για τι υποδομέ, για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιήσει κανείς τα ταμεία συνοχής και τα διασώτικα ταμεία. Άρα λοιπόν χρειάζεται να δούμε πώς μπορούμε ε, να εξασφαλίσουμε άλλα εργαλεία τα οποία θα μας βοηθήσουν στο να επιτύχουμε την απασχόληση, την κοινωνική ε, πρόοδο κτλ. Δηλαδή να κάνουμε ένα είδος συνδυασμού και αυτά να τα δούμε σε συνδυασμό με το επενδυτικό αυτό ταμείο προς την ανάπτυξη. Δηλαδή με το σχέδιο Juncker, για να το πω έτσι όπως συνηθίζουμε να το λέμε, για να μην υπάρχει κάποια σύγχυση. Δηλαδή, το Εύση, που είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα επιπρόσθετο έργο το οποίο θα χρηματοδοτεί ό,τι δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα διαφορετικά ταμεία. Δηλαδή, θέλουμε να φέρουμε συνέργειες, να συντονιζόμαστε καλύτερα, αν για παράδειγμα έχουμε ταμεία συνοχής. Για να χτίσει μια τέτοια είδους αίθουσα, ε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως για την οικοδόμηση και την κατασκευή. Υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Μήπως θα μπορούσαν λοιπόν αυτά τα κονδύλια, και το λέω έτσι για να είναι πιο παραστατικό, να βρεθούν από το εύση Γιατί ο κανονισμός αυτός ε, επιτρέπει να βρεθούν κάποιες συνέργειες χωρίς να χαθούν ε, πουθενά οι στόχοι ούτε των Ταμείων Συνοχής ούτε οι στόχοι του ΕΦΣΗ Δηλαδή Ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι τη ε, πολιτική συνοχή και γι' αυτό είναι και προφανέ ότι όσοι συνέργεια περισσότερο μπορούμε να δημιουργήσουμε τόσο καλύτερα και τόσο πιο πολύ θα πρέπει να την προωθήσουμε. Τώρα, όταν έχουμε επενδυτικέ πλατφόρμε, θα έπρεπε να μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα να έχουμε, για παράδειγμα, ένα έργο το οποίο τη πλατφόρμα αυτό χρηματοδοτείται από το διαστροτικά ταμεία, ένα από το ΕΦΣΥ και θα μπορούσε και ένα κομμάτι αυτή τη πλατφόρμα, ένα δηλαδή υποέργο, Ε, να βρει και κάποιο άλλο ίδιο χρηματοδότηση στη χώρα μου. Γιατί δίνω πάντα το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Έχουμε 150 εκατομμύρια διαρθρωτικών ε, ταμείων για το κοινωνικό ε, κλάδο. Οπότε, τι σημαίνει αυτό. Πως αν θέλουμε αν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε όλα τα φιλόδοξα σχέδια που έχουμε, πρέπει να βρούμε επιπρόσθετα κονδύλια. Άρα λοιπόν εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε στο παιχνίδι τα κονδύλια από το ΕΦΣΥ. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση. Δεν μπορεί το Ταμείο αυτό να υποκαταστήσει την πολιτική συνοχή. Θα μπορούσε όμω να θεωρηθεί ω υποβοηθητικό εργαλείο για την πολιτική συνοχή, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα έργα και να βρούμε τι συνέργειε και το συντονισμό που χρειάζεται. Και γι' αυτό απευθύνω μια έκκληση προς τους εισηγητές έτσι ώστε στον οικονομικό, στον χρηματοδοτικό κανονισμό να λάβουν υπόψη αυτά τα έργα, αυτές τις βελτιώσεις, αυτές τις συνέργειες μέσω ενός καλύτερου συνδυασμού των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ο κύριος Ολμπρίχτ. Euh, euh, euh, Εγώ, Πρόεδρε, θα να σταθώ σε δύο σημεία, σε δύο τροπολογίες που έχουμε. Πρώτα που τα θεωρώ θετική, την τροπολογία, με τον όσων που ο κύριος Φερνάντες, την υπαριθμών 109. Ε, προτείνει να διαγραφεί το να υπάρχει δυνατότητα για πλέον πόρους που θα δοθούν στα κράτη-μέλη. όσον αφορά το έψη και την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. Πολύ εύστοχη αυτή η τροπολογία. που αφορά το, τα κράτη-μέρη τα οποία έχουν τώρα τη δυνατότητα να είναι πιο δυναμικά και δίνει και περισσότερη ευελιξία αλλά να μην είναι δυνατόν να είναι τα δοχεία οι πολιτικές και να παίρνουμε πόρους από τη μία τα πάμε στην άλλη. Όμως, έχουμε στην τροπολίτη υπάρχουν 20 και έχουμε αυτό το αποθεματικό κρίσης για την Ένωση. Αυτό προτάθηκε και μετά καταργήθηκε. Δεν έχουμε τώρα τέτοιο αποθεματικό γιατί η πρόταση απορρίφθηκε. Άρα ο σκοπός του κανονισμού είναι να, να επανεισαγάγει αυτό το αποθεματικό. Θέλετε να το ορίσετε. Πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Κύριος Κέλμελ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια και τον εισηγητή. Πιστεύω ότι δείχνει η μέχρι τώρα δουλειά σας πόσο μεγάλη εμπειρία έχετε ε, και δεν κινείστε καθόλου αφηρημένα, αλλά πολύ συγκεκριμένα με τις προτάσεις σας. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι με οποιοδήποτε μέσο πρόσθετης χρηματοδότησης ε, ή με οποιοδήποτε πρόσθετη αρμοδιότητα αυξάνεται και η πολυπλοκότητα. Είναι προφανές αυτό. Και όταν αυξάνεται η πολυπλοκότητα τότε μειώνεται η διαφάνεια και από μέσα και απ' έξω. Και για τους μέσα δηλαδή και για τους εκτός. Εγώ καταλαβαίνω ε, ότι αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι πολύπλοκο ε, τη πρόσθετη χρηματοδότηση. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι καλό συγκεκριμένα μέτρα να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από διάφορα προγράμματα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και εκεί πραγματικά τίθεται το ερώτημα τελικά. Πετυχαίνουμε τους στόχους όπως τους έχουμε ορίσει. δώσω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και ο συνάδελφος Φερνάντες. Μπορεί να θέλει κάποιος να χρηματοδοτήσει ένα κτίριο. Λογικά αυτό θα πρέπει να θεωρείται ένα μέτρο. Όταν όμως ε, το διασπόμε και το χωρίζουμε σε διάφορα τμήματα. Τελικά έχουμε ένα πρόγραμμα κατακρεματισμένο σε πολλά μέρη και ανάλογα και με το ποιος το χρηματοδοτεί ε, δεν μπορεί να καταλάβεις τελικά τι, στόχοι, ε, τι στόχους επιτυγχάνει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ε, επίσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τα πράγματα. Θέλουμε λοιπόν σαφώς καθορισμένα κριτήρια και μόνο μέσω αυτών και όχι με τελείως διαφορετικά κριτήρια να προχωρούμε. Γιατί επαναλαμβάνω με την ανακατανομή των κονδύλων χάνει τη διαφάνεια. Μπήκαμε λοιπόν και στα πρακτικά θέματα. Σε μια προηγούμενη ζωή, εγώ είχα ζητήσει ευρωπαϊκά κονδύλια και τι κάναμε, βασανίζαμε τα διάφορα έργα που είχαμε έτσι ώστε να καταφέρουμε να τα τσαλακώσουμε μέσα στις δυνατότητες που είχαμε χρηματοδότησης. Γιατί κάθε πρόγραμμα είχε πια μια πολυπλοκότητα η οποία δεν είχε νόημα. Και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι η γραφειοκρατία. Και αυτό θα πρέπει να πατάξουμε με αποτελεσματικότητα. Eh bien, je pense qu'on arrive à Νομίζω όμως ότι φτάσαμε στις 3 παρα 5, φτάσαμε στο τέλος. Δεν ακούσαμε βέβαια το ελεγκτικό συνέδριο εδώ, αλλά επειδή θα ακούσουμε το ελεγκτικό συνέδριο και μετά. Μήπως να σας δώσω το, συνά... το λόγο για να απαντήσετε εσείς στους συναδέλφους αγαπητή συγγήτρια, και μετά θα κλείσουμε αυτό το πρώτο τμήμα γύρω στις 3. Και ίσως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσει, λέει η συγγήτρια. Donc, voulez ah, uh, Υπάρχει ο χρόνος και αν έχουμε προσώπους των πολιτικών ομάδων, ίσως θα μπορούσαν οι δύο ερωτήσεις μου να απαντηθούν. Με τον συνάδελφο Βαντενκάμπα που αναφέρθηκε σε μια πρωτοβουλία. Φυσικά μιλάμε για την προσέλκυση ιδιωτικού κεφαλαίου, αλλά για την ε, ε, διαχείριση. Ε, δεν θέλουμε να υπάρξει περισσότερο διοικητικό άχθος. Ο στόχος είναι το ιδιωτικό κεφάλαιο, επαναλαμβάνω. Για το ΕΦΣΥ Ήταν πολύ αμφιλεγόμενη όλη η συζήτηση που είχαμε στο δημοσιονομικό κανονισμό. Η διατύπωση είναι ΜΕΙ. Έχουμε όμως και τον κανονισμό για τα δραστικά ταμεία. Αν κάνουμε απαλληφή, διαγραφή, είτε δεν κάνουμε, δεν αλλάζει τίποτα, γιατί ο κανονισμός ε, για τα διαρθρωτικά ταμεία είναι αυτός ο οποίος εδώ ε, ισχύει, αυτός που εφαρμόζεται. Δεν έχω προσωπικά κάποια άποψη Απλά νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε. γιατί θα μπορούσαν ακόμη και για τους τίτλους ε, του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου ε, να συγχαίω με κάποια πράγματα και να μην είναι ξεκάθαρο. Εγώ νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να δώσουμε στον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν το λόγο για να απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω δύο λόγια όσον αφορά τη μελέτη επιπτώσεων και τις επικρίσεις σε σχέση με το τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Πρόκειται για μια εργαλειοθήκη. Και βάσει της νομοθεσίας επιλέγονται τα πιο δόκιμα εργαλεία. Βάσει του κανονισμού, οπότε και εμείς θα πρέπει να δούμε το πώς δεν θα γίνει επάπεινο προβληματισμό στο ότι τι θα κάνουμε κάθε πολιτική. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε την επιλογή πιο αποτελεσματικά. Είπαμε ότι από τον προϋπολογισμό που βασίζεται στη δραστηριότητα θα πάμε σε άλλου είδους κριτήρια. Ε, επομένως τα προγράμματα θα έχουν ως στόχους κάποιους δείκτες απόδοσης και επίδοσης. Και αυτό κάθε τόσο συμπληρώνεται από αξιολογήσει. Όμως αυτό δεν θέλουμε να δουλεύει αυτόματα. Ε, είπαμε, οι αποφάσεις είναι πολιτικές, δηλαδή προέρχονται από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Εμείς απλώς ενημερώνουμε τα δύο θεσμικά όργανα. Άρα δεν θέλουμε αυτόματο σύστημα και γι' αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ενημέρωσης περί των επιδόσεων και αποτελεσμάτων και από την άλλη μεριά της θεμητής επιλογής που δικαιούνται να κάνουν τα κρατημέλη και το κοινοβούλιο. Σε αυτή τη βάση αυτά έχω να σχολιάσω. Merci. Monsieur Ο κύριος Ashworth. Θέλει να δώσει κάποιες απαντήσεις στους συναδέλφους. Όχι. Νομίζω ότι όλα τα έχουμε καλύψει. Θα ακούσουμε βέβαια αργότερα και το ελεγκτικό συνέδριο και θα ακούσουμε και τις παρατηρήσεις τους για κάποια από τα σχόλια που έγιναν τώρα. Είναι, ακριβώς τρεις η ώρα. Άρα λοιπόν προτείνω να το κλείσουμε εδώ και να ξεκινήσουμε μάλλον να αφήσουμε εδώ την κοινή συνεδρίαση και να ξεκινήσουμε με την ακρόαση και τις προσωπικότητες οι οποίες θα λάβουν μέρος σε αυτό το εργαστήριο. Ωραία, λοιπόν, για μερικά λεπτά διακόπτουμε τη εργασία μας. Τρεις και πέντε ακριβώς θα ξαναξεκινήσουμε. Et vous pouvez y aller parce que vous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 και με μεγάλη μας χαρά Madame και εγώ τώρα θα διευθύνουμε αυτό το εργαστήρι προβληματισμού και είπαμε ότι θα συστήσουμε αυτήν την απλούστευση του δημοσιονομικού κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποίησε τους καλύτερους εμπειρογνώμονε της ούτως ώστε να συντηθεί και να συνταχθεί ένα κείμενο για αυτό το σκοπό. Οπότε είπαμε να υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών και επίσης θα ακούσουμε τις πρώτες παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Μια γενική έποψη των πραγμάτων, αλλά στη συνέχεια θα ακούσουμε και διάφορους άλλους. Άλλους εμπλεκομένους, οι οποίοι θα μας πούν τις παρατηρήσεις τους, ούτω ώστε να δούμε κατά πόσο αυτή η απλούστευση θα είναι πραγματικά μια απλούστευση σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκομένους στην υπόθεση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Πρόκειται για σειρά ακροάσεων που υπόσχονται πολλά. Κυρία Πρόεδρε, έχετε τη Θέλω να καλωσορίσω όλους τους ομιλητές. Ε, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ελπίζω να μπορέσουμε να ενημερωθούμε για διάφορα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά την χάρη κατάρτιση προπολογισμού βάση ε, επιδόσεων, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, αν μπορείτε κάτι να προσθέσετε έχουμε καλέσει κάποιον, κατά σύμπτωση από το δικό μου σπονδιακό κρατήριο, θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις το αρμόδιο για τα κοινωνικά. Επίσης έχουμε το ΕΦΣΙ και τα διαρθρωτικά ταμεία, είναι ένα θέμα. Έχουμε καλέσει και έναν επιστήμονα που θα μας πει τα σχετικά και στην Περιφερειακή Επιτροπή υπάρχει σχετική ε, εργασία. Θέλουμε να υπάρχει συνεργασία. Είμαστε επικριτικοί σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση κεφαλαίων ε, αναπτυξιακών για άλλους σκοπούς, όμως ε, σε ό,τι αφορά επίσης την εξωτερήκευση Ήθελα να σχολιάσω επίσης την πρόταση που υπάρχει στο κείμενο για τη διαβούλευση ε, με τους πολίτες για τη δημοσιονομικό κανονισμό, τις δημοσιονομικές ε, διατάξεις. Καλό είναι ίσως ε, να δούμε αυτό στην πράξη πώς θα μπορούσε να γίνει. και κάτι που λέει και ο κανονισμός Omnibus για τη σύγκρουση συμφερόντων. Η πρόταση της Κομισιότητας για τα Διαρθωτικά Ταμεία λέει ότι αυτό που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ισχύει και σε επίπεδο κρατών μελών. Έχουμε καλέσει έναν από την Τσεχία για να μας ε, διαφωτίσει από αυτόν Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους ομιλητέ. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως ε, με το ελεγκτικό συνέδριο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λαζάρου που βρίσκεται εδώ, να ευχαριστήσω και το ελεγκτικό συνέδριο, την ομάδα του και ω εισηγήτρια αλλά και ω πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εμπεριστατωμένη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που μας βοήθησε. Πήραμε πολλά τμήματα από αυτήν ε, και μας ε, διευκολύνεται τη ζωή. Σίγουρα ε, θα μπορούσαμε να είχαμε και εμείς καταθέσει περισσότερες τοπολογίες, αλλά τις έχετε καταθέσει πρώτοι εσείς και τις λαμβάνουμε υπόψη. Στις δικές σας προτάσεις βέβαια ε, ο βασικός στόχος είναι η υποστασία των συμφέροντων του Ελληνικού Συνεδρίου. Πάντως έχουμε λάβει υπόψη πολλές από τις δικές σας τροπολογίες. Ε, για κάποιες ε, τροπολογίες μπορεί να μην συμφωνώ απόλυτα. Είμαστε προετοιμασμένοι πάντως να συζητήσουμε και διατεθειμένοι να συζητήσουμε όλες τις τροπολογίες. Κύριε Λαζάρου, παρακαλώ έχετε το λόγο. Mr. Κύριε Αρτουή, κυρία Γκρέσλερ, κύριε Άσουαρτ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συνεισφέρω σε αυτή την ε, ομίγυρη και νομίζω πως η πρόταση που σας κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν φιλόδοξη για την αναθεώρηση του ε, χρηματοδοτικού κανονισμού. Είναι τεράστιο το έργο σας στην αξιολόγηση αυτή της ε, πρότασης και σήμερα καλύπτουμε μια σειρά από τα θέματα τα οποία πρέπει να καλύψουμε Ξέρετε, επειδή εμείς ε, καταθέτουμε τη γνώμη μας, τη γνωμοδότησή μας, πόσο δύσκολο είναι να περάσει κανείς από 900 σελίδες τροποποιημένο νομικό κείμενο και τις συνημένες εξηγήσει του προτινόμενου ε, κανονισμού και της ε, τροποποίησης αυτής. Θα εστιάσω σε τρία σημαντικά κομμάτια της γνωμοδότησής μας, και μετά εντάχει θα ασχοληθώ με τρία άλλα θέματα πριν κλείσω με ένα αίτημα να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε. Το πρώτο κομβικό σημείο έχει να κάνει η ανάγκη μίας ενιαίας ανα, αναφοράς για τη λογοδεσία και την αποτελεσματικότητα. Και νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υποβολή αναφορών δεν μας έχει πει αν απλώς τον ίδιο χρόνο θα ε, δημοσιεύει την υφιστάμενη έκθεση ή αν θα έχουμε μία άλλου είδους έκθεση στην περίπτωση αυτή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη, ε, λαμβάνοντας υπόψη την, ε, τις συστάσεις δικές μας ε, για τη διακυβέρνηση. Το να κάνουμε κάτι τέτοιο θα φέρει στη σύγχρονη εποχή την αναφορά που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει δείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως ανοιχτεί στην αλλαγή με το πακέτο για την ολοκληρωμένη οικονομική αναφορά και το γεγονός πως αποφάσισε να το εντάξει στις προσπάθειες που κάνει, αλλά δεν φτάνει αυτό αρκετά μακριά. Γιατί χρειαζόμαστε μία ενιαία έκθεση ε, λογοδοσίας, η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς πρακτικές, τις βέλτιστες πρακτικές. Και θα πρέπει αυτή να συμπεριλαμβάνει πρώτα απ' όλα της Προεδρίας, σύνοψη δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων για κάθε χρονιά, συζήτηση των κινδύνων με την ε, δήλωση διακυβέρνησης και το γεγονός και το πώς ε, ελέγχει την κατάσταση. Επίσης, η η έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής για το πλήσον των εξωτερικών μελών. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συνοδεύουν τα παραδοσιακά κομμάτια των οικονομικών λογαριασμών, οι οποίοι θα πρέπει να συνοδεύονται από μία δήλωση μέσω μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας και όλα αυτά θα πρέπει να κατα, ε, τα θα σε εμά ε, σε κατάλληλο χρόνο για τον έλεγχο των λογαριασμών και για ελέγχους συνέπειας και συνοχής έτσι ώστε να μπορούμε εμείς την ανεξάρτητη γνώμη μας να την καταθέτουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής. Το δεύτερο κομβικό σημείο είναι να προχωρήσουμε ε, ε, στην εφαρμογή του προπολογισμού που θα βασίζεται στην αποτελεσματικότητα. Δηλαδή θα πρέπει η αιρεσιμότητα να είναι αποδοτικότητα και όχι κοστολόγηση. Και εδώ έχουμε παρουσιάσει παρατηρήσει για το πώ θέλει να το επιτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στηρίζουμε την κίνηση αυτή οι πληρωμές να γίνονται για τα ε, ε, αποτελέσματα τα οποία έχουν επιτευχθεί σε όλη την γάμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού και καλωσορίζουμε τις προσπάθειες να απλουστεύσουμε ε, κάποιους, κάποιες διευθετήσεις πληρωμής οι οποίες είναι υπέρ των δύο περίπλοκες. Η εξηγήση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει πως η stand-by λύση που είναι κερδοφόρα project μέσω χρηματοδοτικών οργανισμών σημαίνει πως αν πως εγκαταλείπουμε την αρχή του μη κερδοφορία, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να στηρίζουμε. Επίση, η εθελοντική εργασία μα λέει πω θα πρέπει να κοστολογείται τη στιγμή τη απόφαση χρηματοδότηση. Κατά τη γνώμη μα, αυτό αυξάνει τον κίνδυνο μη επιλέξιμων δαπανών και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Το τρίτο κομβικό είναι η ευθυγράμμιση των διαδικασιών απόφαση και σύνταξη προπολογισμού. Δηλαδή, θα πρέπει στην πρόταση που, έχουμε κάνει, που έχουμε πολλές ε, αλλαγές ε, καταλήγουμε σε ένα σχήμα αρκετά περίπλοκο με επιπλέον εξαιρέσεις ε, στις διάφορες αρχές που έχουμε ήδη βάλει. Είπαμε η μεταφορά θα πρέπει να γίνει από τη διαμοιρασμό ευθύνης χήνης να γίνει σε ένα σύστημα όπου την απόλυτη ευθύνη θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε επίσης και για το θέμα της μεταφοράς κονδυλίων από το ένα έτος στο άλλο, κάτι το οποίο το carry over δηλαδή που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Το ίδιο συμβαίνει και για τις εσωτερικές αποδόσεις. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής αυξάνει τον αριθμό κατηγοριών ε, και επιτρέπει αυτές οι αποδόσεις να χρησιμοποιούνται και για άλλου στόχου από αυτού για τον οποίο αρχικά είχαν ε, στοχοθετηθεί αυτό γίνεται με λογιστικό τρόπο και έχουμε αυτή τη μεταφορά από εσωτερικές αποδόσεις σε γενικές αποδόσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για παράδειγμα. Στον προϋπολογισμό του 2017 είχαμε μείωση των ανάληψων υποχρεώσεων για την άμεση επιδότηση ε, στους γεωργούς κατά τρία δις έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η εσωτερική απόδοση από τις οικονομικές κυρώσεις. Έχουμε πει λοιπόν ότι οι άμεσες επιδοτήσεις θα πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνες και να ληφθούν υπόψη και αυτά τα 2,3 των καταλογισμών να θεωρηθούν γενικά έσοδο του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Ξέρετε πω αυτά τα τρία κομβικά ζητήματα δεν είναι τα μόνα τα οποία συζητάμε στην δική μα γνωμοδότηση. Θα τονίσω άλλα τρία. Καταρχήν, είναι πολύ θετική η πρόταση για την οικονομική χρηματική παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά εκεί θα πρέπει να μα ξεκαθαρίσει τι ακριβώ προτείνει και τι θέλει να πετύχει. Για παράδειγμα, πώς ε, οι κοινέ διατάξεις θα, θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα ε, ε, υπολογίζουμε την αποδοτικότητα. Δεύτερον, ο συνδυασμός διαφόρων ε, χρηματοδοτικών εργαλείων από πολλά διαφορετικά κομμάτια του κανονισμού. Αυτό μοιάζει να είναι ε, αντίθετο με την αρχή της απλούστευσης. Η δική μας σύσταση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει δικλείδες ασφαλείας που θα είναι αρκετές έτσι ώστε τέτοιου είδους συνδυασμός να ε, σέβονται τους κανόνες για τις κρατικές επιδοτήσεις και για ε, την ε, ε, για τα κονδύλια ε, και τον τρόπο πληρωμή αυτών. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά νωρί για κάποια ε, χρηματοδότηση εξωτερικής δράσης ε, αυτή η διάταξη, γιατί πολλέ φορέ η αξιολόγηση δεν έχει φτάσει στην ώρα τη και δεν γίνεται να επεκτείνουμε με τον τρόπο που προτείνεται. Και τέλο, βοηθήστε μα να σα βοηθήσουμε. Είμαστε ο εξωτερικό ελεγκτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε εσωτερικό όργανο. Και έχουμε σκοπό εδώ εμεί να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο και, και προετοιμάζουμε την έκθεσή μας και την παρουσιάσουμε. Εμείς δεν θέλουμε και διαφωνούμε με το να προαποφασίζεται πώς, ε, ε, τι μορφή θα έχει η εκθεσή μας. Γιατί έχουμε και τις ειδικές εκθέσεις και αντί να μας ενδιαφέρει πιο πολύ το φορμάτι της έκθεσής μας, θα πρέπει ο οικονομικός κανονισμός να επιτρέπει σε εμάς να αποφασίσουμε πώς θα τα ε, διατυπώσουμε και τι, τι layout θα έχουμε. Και γι' αυτό η τροπολογία 208 μας δημιουργεί ανησυχίες. Πριν κλείσω, θα ήθελα να αντιμετωπίσω ε, την ερώτηση του κυρίου Σαβαρμά από λίγο προηγουμένως. Γιατί δεν υπάρχει δηλαδή ο ορισμός των αποτελεσμάτων. Εμείς είπαμε στην δική μας γνωμοδότηση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει, την, αλλάζει την αρχή της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και λέει χρηστή οικονομική διαχείριση και αποτελέσματα. Όμως δεν δίνουν έναν ορισμό του τι ακριβώς σημαίνει απόδοση αποδοτικότητα. Και στις συστάσεις τις δικές μας τους καλούμε να παρουσιάσουν και ένα τέτοιο ορισμό. Θα αναφερθώ τώρα στην ετήσια έκθεση του 2015, όπου στο κεφάλαιο 3 μιλάμε για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και εκεί δώσαμε έναν ορισμό της αποδοτικότητας υπό τους τέσσερις πυλώνες που είναι το input, output, αποτελέσματα και συνέπειες. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά είναι τα τέσσερα σημεία αυτά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρουσιάσει έναν ορισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ των διαφόρων ελεγκτικών αρχών σε όλη την αλυσίδα της λογοδοσίας να γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει αποδοτικότητα και να υπάρχει ένας κοινό τρόπος μέτρησης αυτών των αποδοτικότητας με ε, δείκτες αποδοτικότητας που θα εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο καθ' όλη τη διαδρομή. Κυρία Γλέσσερ. Κύριε Αρτουή, κύριε Άσουαρτ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμείς είμαστε δεσμεσμένοι στο να σας βοηθήσουμε, στο να ασκείτε τα ελεγκτικά σας καθήκοντα. Εμείς στη γνωμοδότησή μας για την αναθεώρηση του ε, κανονισμού αυτού ε, τονίζουμε κάποια θέματα τα οποία εσείς θα πρέπει να δείτε και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ανταλλαγή euh, Ευχαριστούμε κύριε Λαζάρου για τις παρατηρήσεις σας. Για το ότι ήρθατε για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση τώρα. Όσον αφορά αυτού του είδους τα έσοδα ειδικού προορισμού, μήπως θα πρέπει γενικότερα να δούμε ανοφελεί αυτή η πρακτική η οποία κυριαρχεί όσον αφορά τα λογιστικά, τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, για αυτά τα ειδικό προορισμό. Είπαμε σήμερα ότι θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειε βάρο του Δικαστήριου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καθυστέρηση λήψη αποφάσεων και πρόκειται για αυτή την αποζημίωση, αυτή την χρηματική ποινή από κάποιους ειδικού πόρους που πάνε κατευθείαν στα κράτη-μέλη. Όμως, όποτε υπάρχει κάποια τέτοια επιβολή χρηματικής ποινής, αυτή επιβαρύνει τον κοινωτικό προπολογισμό. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου είδους έσοδα ειδικού προορισμού για κάποια έσοδα που αφορούν χρηματικές ποινές. we διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν βασιμοί λόγοι, ούτως ώστε να έχουμε εξωτερικά εσωτερικού προορισμού, διότι τα κράτη-μέλη τα οποία εισφέρουν σχετικώς θέλουν αυτοί οι πόροι να αξιοποιηθούν σε συγκεκριμένο τομέα. Φέρει το έρασμος. Όμως, δεν μαθαίνουμε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι τόσο ώστε να έχουμε κάποιο είδου εσωτερικά εσωτερικού προορισμού και να μην να μην γίνονται να μην θεωρούνται, συγγνώμη, μέρος του γενικότερου προπολογισμού οι διορθώσεις του γεωργικού προπολογισμού. Θα πρέπει η αρχή του προπολογισμού να έχει λόγο στο πώς θα δαπανηθούν αυτοί οι πόροι, πώς θα γίνει ο καταλογισμός, διότι ε, έτσι, έτσι φροντίζουμε αυτά τα εσωτερικά εσωτερικού προορισμού. Κύριε Φεραντές, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το Ταμείο Βοηθείας για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, χρησιμοποίησαμε αυτό το μοντέλο, αυτό το πρότυπο του εξ, των εξωτερικών εσόδων προορισμού, ούτω ώστε να υποχρεώσουμε εντό εισαγωγικών τα κρατημέλη να τηρήσουν αυτή την υποχρέωση της συνεισφοράς και με αυτόν τον τρόπο είπαμε ότι θα υπάρχει αυτό το καταπίστευμα και θα υπόκειται σε έναν έλεγχο της απαλλαγής. Ερωτώ, τι δυνατότητες υπάρχουν ούτως ώστε αυτό το ταμείο να υπάρχει χωρίς να υπάρχει και καταπίστευμα κάποιου είδου δηλαδή εξωτερικά εξωτερικού προορισμού. Πώς θα γινόταν αυτό, τι λύση θα δίνονταν γιατί τα κράτη-μέλη διερευνούν, σκέπτονται κάποια λύση, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για το ηλεκτρικό συνέδριο. Δηλαδή να υπάρχει ένα πλαφόν, μια οροφή και ε, να μην ξεπερνάμε αυτή την οροφή με, το, με, το, με τα εξωτερικά έσοδα προορισμού. Είπαμε μέχρι εκεί, τέλος. Υπάρχει αυτό το πλαφόν. Αν όμως πρόκειται για γενικού είδους δαπάνη, συνήθεια δαπάνη, ε, τότε μπορεί να ξεπεράσουμε το πλαφόν και θα πούν τα κράτη-μέλη όχι, μια που περάσαμε το πλαφόν δεν δίνουμε λεφτά. Άρα πώς θα μπορούσαμε να βρούμε μια άλλη λύση. Γιατί ούτε εμένα μου αρέσει αυτό το εξωτερικό έσοδο ειδικού προορισμού. Αλλά είπαμε ότι μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε λύση που να μην είναι καθαρά διακυβερνητικό χαρακτήρα αλλά να μπορούμε να έχουμε έλεγχο επί του πώς δαπανώνται τα χρήματα. Άρα για να το δούμε. Γιατί τότε η εναλλακτική θα ήταν κάποιο είδου ε, ταμείο, καταπίστευμα τέλο πάντων, διακυβερνητικό μεταξύ των κρατών μελών. Τι λέτε. Τι είναι που να έχουμε, για... έχουμε να διέξουμε μεταξύ κάποιου πράγματος που είναι κακό και άλλου πράγματος που είναι πολύ κακό. Τι θα διαλέξουμε. Το κακό και το χειρότερο, λέει ο Λαζάρο. Σας διευκρινίσω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όσον αφορά το εξωτερικό εσωτερικού προορισμού ή αυτού του είδους τα εξωτερικά καταπιστεύματα. Αυτά τα ταμεία. Απλώς σταθήκαμε στο θέμα των εσωτερικών εσωτερικού προορισμού και σας εξηγήσαμε γιατί κατά τη γνώμη μας δεν το εγκρίνουμε, δεν το υποστηρίζουμε. Διότι αυτό αντιβαίνει στην ε, διαφάνεια, δεν παρέχει την ευκαιρία στο Κοινοβούλιο να έχει λόγο σε σχέση με το πώς θα δαπανηθούν αυτοί οι πόροι. Οπότε όλα τα έσοδα εγγράφονται στα έσοδα και όλες οι δαπάνες στις δαπάνες. Αυτή είναι λοιπόν η αρχή της καθολικότητας και της ενότητας του προπολογισμού. Τώρα για τα καταπιστεύματα να σας πω πως είναι κάποιο είδους ιδιάζοντα ταμεία που δεν συνεισφέρουν στην ειλικρίνεια και την τιμιότητα των δημόσιων λογαριασμών. Τώρα η γνώμη σας για όλα αυτά κύριε Λαζάρου είναι η γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου. Euh, για το ελεγκτικό, για, το, για την απλούστευση, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας. Πιστεύετε και επιβεβαιώνετε την εκτίμηση ε, την, ε, που κάνουμε. Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να τελειοποιηθεί ακόμα πολύ πιο πολύ και πως δεν έχει πετύχει τους στόχους της και επίσης αυτή η απλούστευση θα μπορούσε να έχει και κάποιες αρνητικές συνέπειες. Uh, Ευχαριστώ πολύ το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε μέσω της γνωμοδότησής μας. The commission proposal... Είναι ότι η πρόταση της Κομισιόν ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν φτάνει αρκετά μακριά. Δηλαδή δίνει μια σειρά από εξαιρέσεις οι οποίες περιπλέκουν ε, την κατάσταση και προσθέτουν ε, περίπλοκες διατάσεις, διατάξεις χωρίς να οδηγούν σε μεγαλύτερη απλούστευση. Οπότε είναι με βήμα προς την κατεύθυνση, αλλά πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Ωραία λοιπόν. Θα καλέσουμε τώρα τον κύριο Ματίας Μπολ, Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης από το κρατήδιο της Βάδης Βερτεμβέργης. Κυρίε Κυρίες και κύριοι, με τιμά ιδιαίτερα, Δόκτωρα Κρέσλε, κυρία του, κυρία Σχόρφ, μου δίνει τη δυνατότητα σήμερα να να μιλάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Με τιμά λοιπόν ιδιαίτερα, δόκτωρα Γκρέσλε, κύριε Του, κύριε Άσφορτ, να το που να είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω την προοπτική μιας διαχειριστικής αρχής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στην Βάδη ε, ε, έχουμε ένα μικρό πρόγραμμα, επιχειρησιακό πρόγραμμα 260 εκατομμυρίων ευρώ, οι βασικές κοινωνικές δαπάνες βέβαια πραγματοποιούνται από άλλους οργανισμούς. Παρ' όλα αυτά το ΙΣΕΦ e είναι σημαντικό και το χρησιμοποιούμε κυρίως για τον έλεγχο και την ανάπτυξη νέων εργαλείων, για την καταπολέμηση, παραδείγματα, της μακροχρόνιας ανεργίας. Τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετές επιτυχίες, πολλά μέσα χρηματοδοτήθηκαν από άλλους οργανισμούς μετά την εκπνοή της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΚΤ. Τώρα, ποια είναι οι πρακτικές προκλήσεις για μια διχειριστική αρχή σε ό,τι αφορά την κατάσταση προβλησμού βάση επιδόσεων. Όσο πιο καινοτόμο είναι ένα μέσο, τόσο πιο δύσκολο είναι να προβληθεί οι επιδόσεις, ε, το output αυτού του εργαλείου. Έχουμε διάφορες εξελίξεις όπως την αγορά εργασίας για παράδειγμα που είναι πολύ δύσκολο ίσως και αδύνατο να εκτιμήσει κανείς 7 χρόνια νωρίτερα. Οι ε, αλλαγές επίσης ε, του επιχειρησιακού προγράμματος για την εντόπιση νέου, ε, μιας νέας κατάστασης είναι κάτι στη θεωρία εφικτό, αλλά στην πράξη δημιουργεί προβλήματα. Υψηλότερο το κατόφλι και μεγαλύτερε ανάγκε και σε προσωπικό κτλ. Ένα καθόδη ζήτημα είναι ότι αυτή η κατάρτιση προπροσμού βάση επιδόσεων που επιβάλλεται από τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις ε, φέρνει κάποια αποτελέσματα. Θα πρέπει, παραδείγματο χάρη, διχειριστικέ αρχέ να μην παίρνουν ρίσκα και θα πρέπει να εστιάζει η παρέμβαση του ΕΚΤΑ σε εύκολα προβλέψιμους τομείς, ε, σε πιο αξιόπιστα προβλέψεις. Βέβαια, Πρέπει να δούμε κατά πόσον οι τομείς αυτοί είναι και πλέον αναγκαίοι ή ευκταίοι για κάθε κράτος μέλος. Υπάρχει ένας κίνδυνος, κίνδυνος του λεγόμενου creaming effect, δηλαδή οι παρεμβάσεις να εστιάζουν μόνο σε ομάδες ε, ανθρώπων που υπόσχονται γρήγορη και μετρήσιμη επιτυχία. Δηλαδή τελικά τι κάνουμε, ενισχύουμε τους ισχυρούς και τους άλλους τους ξεχνάμε. Για να σας ένα παράδειγμα. Η ομάδα μακροχρόνια ανέργων δεν είναι καθόλου μεγενής. Κάποιοι από αυτούς είναι πολύ κοντά στην αγορά εργασίας, άλλοι είναι πολύ μακριά και έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά πολύπλοκα προβλήματα ε, με την ψυχική του υγεία, για παράδειγμα, μπορεί να τοξικομανείς κτλ. με βάση μάλλον τον κανόνα ε, της ε, το performance-based budgeting εστιάζει το έκτα στους μακροχρόνιους νέου που είναι πιο κοντά στην αγορά εργασίας και όχι που χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια για να βρουν δουλειά. Α πάμε σε ένα δεύτερο καρθόδε ζήτημα. Ω διαχειριστική αρχή θα πρέπει να δεις τι θα κάνεις αν δεν επιτύχεις τους στόχους σου πρέπει να προτιμάς ε, εργαλεία που είναι δοκιμασμένα, που θα έχουν επιτυχία. Και εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κοινωνική καινοτομία που θα πει πειραματισμός, ανάπτυξη νέων εργαλείων και μέσα για την αντιμετώπιση ε, της, ε, των κοινωνικών προβλημάτων. Έχουμε και το άρθρο 9 του κανονισμού που λέει ότι έχουμε καθήκον Προ την κοινωνική καινοτομία. Στην χειριστική αρχή επίση θα πρέπει να δούμε και τους δικαιούχους. Ούτε αυτοί πρέπει να παίρνουν ρίσκα. ε, πρόκειται για μη κυβερνητικούς, μη κρατικούς κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ε, δηλαδή φιλανθρωπικά ιδρύματα, παραδείγματος χάρη, φιλανθρωπικές ΜΚΟ. Με μικρό δημοσιομικό μαξιλάρι θα έλεγα και ε, δεν έχουν ε, μεγάλες δυνατότητες γιατί μπορούν να, να, αντιμετωπίσουμε και τον κίνδυνο της πτώχευσης. Και το ΕΚΤΑ δεν είναι τόσο ελκυστικό γιατί η γραφειοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παραμένει άλυτο. Και για να ολοκληρώσω, transforms into compliance η επιβολή αυτής της κατάστασης προπολογισμού βάσει ε, της ε, επίδοσης με τη χρηματοοικονομική μόχλευση από εκεί και ε, αποκτά τη δική της δυναμική στη συνέχεια. Επίσης, πολλές φορές οι επιδόσεις γίνονται συμμόρφωση, υπάρχουν άλλοι παράγοντες που δεν λαμβάνονται τόσο υπόψη όσο το πρωτοπόρο πνεύμα κτλ. Υπάρχουν ε, υπάρχει προτίμηση σε δοκιμασμένα εργαλεία και όχι σε νέες προσεγγίσεις που επειδή με κινδύνους ε, και επίσης υπάρχουν και δομικά μειονεκτήματα για ανθρώπους με πολύ κοινωνικά προβλήματα. Ευχαριστώ. Κυρία Γκρέσλη. τελικά δεν ξέρω πραγματικά ε, τι πρέπει να στηρίξουμε, τα βασικά ή αυτούς που έχουν ε, την τόλμη να προωθήσουν ε, κάτι καινούριο, να καινοτομήσουν. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Καταπολέμηση νεανικής ανεργίας. Έχουμε δαπανίσει δισεκατομμύρια για αυτό το θέμα. Τι πετύχαμε, δεν ξέρουμε τι πετύχαμε, γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής έκθεσης και δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία. Τι θα μας συμβουλεύατε, τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, από τη πλευρά των διχειριστικών αρχών του ΕΚΤΑ καλό θα ήταν να μην ρυθμίζονται τα πάντα με βάση τη αρχής ε, της κατάσταση προπολογισμού βάση επιδόσεων, να αφήνεται περιθώριο δηλαδή, να δοκιμαστούν νέα μέσα, να υπάρχει δυνατότητα πειραματισμού. Αλλά να μην φοβάται αυτός που πειραματίζεται ότι θα έχει χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, ε, ουσιαστικά η γοητεία, αν θέλετε, του έκτη είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα πειραματισμού και καινοτομίας. Ευχαριστώ, συνάδελφος Φερνάντες, παρακαλώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Φερνάντες. Εγώ θα μείνω στο θέμα συντονισμού μεταξύ των χρηματοοικονομικών ε, εργαλείων και των ε, διορθωτικών ταμείων. Πρόκειται για κοινωνική κοινοτομία, οπότε και χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά αυτά τα χρηματονομικά εργαλεία. Βάζει τέτοιο πρόγραμμα. Προκειμένου συζητούμε για τη δική σα περιφέρεια, ευχαριστούμε για όσα μα είπατε. Οπότε, αν κάνουμε ένα τέτοιο συντονισμό μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, των Διευθυντικών Ταμείων και των ε, ε εργαλείων, τι θα γίνει. Πώ θα πάει το πράγμα. Εάν δεν κάνετε αυτόν τον συντονισμό, θεωρείτε ότι πρόκειται για καλή ιδέα. Είναι δυνατόν να έχουμε συνέργεια. Γιατί νομίζω ότι η κοινωνική καινοτομία πρέπει και δύναται να συσχετιστεί με αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία όπως το ΆΖΙ. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο το ανέφερε και η εισηγήτρια και η πρόεδρος. Για φακέλους οπότε ε, επικαλούμεθα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τι μπορεί να γίνει τόσο ώστε να έχουμε προγνωστικά των αποτελεσμάτων. Μήπως μπορεί το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Σύνδεσμο να μας βοηθήσει από αυτού. Πότε μπορούμε να μιλούμε για επιδόσεις, για αποτελέσματα όσον αφορά την, την αξιοποίηση των ταμείων όπως αυτά. Γιατί πάντοτε είναι πάρα πολύ ωραία να λέμε για ε, προπολογισμό που έχει να κάνει με τα αποτελέσματα αλλά για να είμαστε τελικά αποτελεσματικοί θα πρέπει να, έχουμε, να το αποδείξουμε έχοντα τα, τα αποτελέσματα. Είναι εδώ να κάνει κανεί προγνωστικά μετά το match. Εύκολο θα ήταν αυτό. Γιατί θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε κάποια ε, αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή να έχουμε νωρίτερα πολύ αισιόδοξο και να πούμε ότι να, ήταν εξαιρετικά τα αποτελέσματα, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και ότι ο ήταν πολύ χαμηλά. Επομένως έτσι έχουμε στρέβλωση. Άρα το, τώρα το θέμα είναι το πώς θα αντιμετωπίσω αυτά τα δύο θέματα. Και η, δε, δεύτερη ερώτηση που είπα είναι το πώς μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο προϋπολογισμό performance based και εν μια εκτέλεση που να βασίζεται στα αποτελέσματα την ίδια σειρά και ακολουθώντας το ίδιο πνεύμα, μήπως τελικά κάνουμε υπερβολικά πολλά με αυτόν τον κανονισμό, γιατί περί τίνος πρόκειται. Συμφωνίες. Συμφωνίες στις οποίες καταλήγουν, έχουμε τα κράτη-μέλη που συνεισφέρουν, είναι μια πράξη αλληλεγγύης. Κάποια κράτη λοιπόν συνεισφέρουν πολύ, και λαμβάνουν κάπως λιγότερα, αντίθετα κάποιοι άλλοι λαμβάνουν παραπάνω από ό,τι έχουν συνεισφέρει. Αυτό είναι η αλληλεγγύη. Είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε από έναν τόσο περίπλοκο κανονισμό που στο κάτω-κάτω ε, καίει την κατάσταση γιατί Πώς μπορούμε να ε, κάνουμε πειράματα για να βρούμε την κατάλληλη λύση όταν όλα ρυθμίζονται με κανόνες. Δηλαδή έχουμε ας πούμε ε, για τη μαθητεία ένα πειραματικό project. Έχουμε κάποιες διαδικασίες που δεν μας επιτρέπουν να μην κάνουμε τίποτα. Δηλαδή το να είναι κανείς καινοτόμος χρειάζεται ένα ελαφρύ πλαίσιο που θα σε επιτρέψει να δείτε ποιε είναι οι καλύτερες λύσεις, τι θα μπορέσετε να δοκιμάσετε και δεν πληρώνει η Ευρώπη στο 100% έτσι κι αλλιώς τι τις αυτέ. αυτές και νομίζω ότι το γεγονός που συνεισφέρει και ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος είναι η καλύτερη εξασφάλιση πως δεν θα πετάξουν τα λεφτά τους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αν το δει κανεί επί τόπου, μπορεί τελικά να καταλήξει να βλέπει σχήματα τα οποία ουσιαστικά είναι καρικατούρα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, κύριε Μπόλ, σας ευχαριστώ για μια πάρα πολύ σαφή και κατανοητή παρουσίαση. Uh, Μην ξεχνάμε λοιπόν πως όλα αυτά τα έχετε δει υπό το πρίσμα του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρέπει βεβαίως να αποφεύγουμε να είμαστε ιδιαίτερα απλουστευτικοί στις αποφάσεις που παίρνουμε. Δεν χρειάζεται υπεραπλουστευμένες λύσεις. Και να μετράμε βέβαια τις συνέπειες, ε, όχι μόνο εκεί, αλλά παράλληλα να προσέχουμε, γιατί εγώ δεν θα ήθελα καν να φανταστώ πως θα παραιτηθούμε από την προσπάθεια για να βρούμε τα βέλτιστα κριτήρια για αποτελέσματα και συνέπειες σε χώρους όπου γίνεται. Και να μην πούμε ότι απλώς ότι δημιουργούμε ουσιαστικά μία φούσκα με τη δική της δυναμική, είναι μία υπεραπλούστευση ή τέλος πάντων πολύ γενικευμένο αυτό που λένε. Θα πρέπει να δούμε πως υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και μπορούν στις διαφορετικές αυτές ανάγκες να εφαρμόσουμε διαφορετικά κριτήρια. Ο κύριο Κέλμελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον Δόκτωρα Μπολ ε, για την παρουσίασή του. Συμφωνώ με τους προλαλήσατε σε πολλά σημεία. Θα ήθελα να εμβαθύνω σε ένα σημείο. δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να καταπιαστούμε με κάτι επειδή είναι δύσκολο και επειδή είναι πολύ πλοκό. Ούτε ε, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν τα πάντα και στη Γερμανία έχουμε εμπειρία που δείχνει ότι κάποιες φορές υπάρχουν ε, τρελές αιτιολογήσεις ε, για διάφορα καθήκοντα ή έργα που δεν έχει κανένα νόημα τελικά να εφαρμοστούν. Και να μην αναφέρω και την αύξηση της γραφειοκρατίας που είναι τελώς αχρίαστη. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι να έχουμε επιτυχημένη εφαρμογή σε διάφορους τομείς. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, αυτήν την, τον ορισμό και αυτήν την αρχή της αλληλεγγύης, για μένα αυτό σημαίνει βοήθεια. Αλλά δεν είναι απαραίτητα ε, σαφές ότι μπορούμε να ορίσουμε με τρίσιμους στόχους για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ουσιαστικά εστιάζουμε σε ένα τομέα και παρέχουμε βοήθεια. Αυτό θα πει αλληλεγγύη. Και φυσικά και χρειαζόμαστε Ευρώπη, ε, στην Ευρώπη αλληλεγγύη, ίσως πολύ περισσότερα από ό,τι μέχρι τώρα. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Και η προσέγγιση είναι πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει να δούμε τελικά ποιος χρειάζεται αλληλεγγύη. Έχω ξανακάνει την πρόταση και στο παρελθόν. Να συζητήσουμε ξεκάθαρα και ανοιχτά κατά πόσον ε, οι καθαρείς φορείς θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερα ποσά τα οποία τα ξαναπαίρνουν στη συνέχεια πίσω. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε πολύ καλύτερα τα προβλήματα αν μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τα πράγματα όσο πιο κοντά στο επίπεδο που παρουσιάζονται, που ανακύπτουν. Εμεί είμαστε ένα ομοσπονδιακό κράτο. Στη Γερμανία έχουμε ομοσπονδιακά κρατήρια, στη δική μου την ε, ε, περιοχή έχουμε την ε, κυβέρνηση τη Στουτκάρδη, από εκεί είναι και ο κύριο Μπολ. Και φυσικά και εμεί ξέρουμε πολύ καλύτερα τα προβλήματα τη ε, Βάδη τα ξέρει και η κυρία Γκρέσλε βέβαια, σε σχέση με την κυβέρνησή μα, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Βερολίνο ή ε, βέβαια και το Βερολίνο ξέρει καλύτερα τα πράγματα από ότι οι Βρυξέλλες. Να στέλνουμε λοιπόν χρήματα εδώ στις Βρυξέλλες και να τα ξαναγυρίζουμε μετά πίσω. Και έχουμε και 28 κράτη-μέλη. Καταλαβαίνετε πόσο πολύπλοκο είναι όλο αυτό. Μπορεί να μην είναι πολύ δημοφιλέσα. Ίσως είναι λίγο γραμμή της Μάρκετ Θάτσερ αλλά νομίζω ότι πρέπει να το, ε, να το συζητήσουμε ξεκάθαρα και ανοιχτά. Και παραλαμβάνω. Εγώ δεν λέω να μειώσουμε τα ποσά για τη Γερμανία. Απλά λέω, επειδή είναι καθαρό σε η Γερμανία και συνσφέρει σε μια ευρώ, ευρύθμος λειτουργούσα ένωση, αλλά νομίζω ότι αν είναι πιο απλή, ε, πιο απλές οι διαδικασίες και οι δομές, θα λειτουργεί ακόμα πιο ευρύθμος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ θετικό το ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί μας έχουν τόσο πολύ καιρό απασχολήσει τα θέματα τα σχετικά με τον προϋπολογισμό και τις επιδόσεις. Επομένω αξίζει να ασχοληθεί κανεί με αυτό που τώρα μα απασχολεί. Πάντω, έχω να πει ότι το performance budgeting και η απλούστευση είναι δύο πράγματα που είναι αντιφατικά μεταξύ του γιατί έχουμε τους παράγοντες της, ε, ε, ε τον παράγοντα κάνει τη ζωή μας ευκολότερη, αλλά την άλλη μεριά έχουμε το θέμα αυτό του performance based budget και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα μετρήσιμα για κάποια ζητήματα τα οποία είναι ε, ποσοτικά μετρήσιμα αλλά πώς κανείς θα διαχειριστεί τα θέματα της ποιότητας και το τρίτο που θα σας αναφέρω είναι ότι στο δημόσιο τομέα που έχω κάποια εμπειρία υπάρχει ένας κίνδυνος που ελοχεύει. Ότι δηλαδή να κυριαρχίζει αυτή η κουλτούρα ε, των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων. Και τελικά να ακολουθεί ο κάθε φορέας, ο καθένας, την πιο εύκολη λύση. Και να μην κάνει αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνει που είναι πιο δύσκολα. Οπότε, ε, τελικά προς τα εκεί πηγαίνουμε, προς αυτή την κουλτούρα των επιδόσεων που δεν είναι αναγκαστικά αυτό το οποίο επιδιώκουμε. Άρα έχω αυτές τις τρεις επιφυλάξεις. Ναι, ναι, ναι, για όλα αυτά, τα, για τους δείκτες, τα στοιχεία, ε, θα πρέπει κανείς να δυσπιστεί. Αυτό έχει να κάνει και με τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Σαραβαμά. Τα συζητήσαμε και στην προηγούμενη συνάντηση αυτά, αλλά για όσους δεν ήταν παρόντες, σας επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είχα πει τότε ότι για αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει πολύ προσεκτικά να ασχοληθούμε με τους ορισμούς και τελικά μην ακολουθούμε την πιο εύκολη λύση και να πέσουμε στην παγίδα που μας ε, περίγραψε ο κύριος Μπόλ. Να δούμε μόνος πώς μπορούμε να προσπάσουμε τα καλύτερα αποτελέσματα με τα δαπανόμενα χρήματα. Ευχαριστώ πολύ. Μία σύντομη παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Κέλμελ, που μου θύμισε κάτι. Έχουμε το εξή πρόβλημα σήμερα. Οι καθαρείς φορείς παίρνουν τμήμα των χρημάτων τους, ε, εφόσον δεν έχουν ε, εκταμιευθεί πλήρως, τα παίρνουν πίσω. Φυσικά λοιπόν και έχουν το συμφέρον να μην ε, χρησιμοποιηθούν ε, οι πιστό στο έπακρο. Ίσως θα ήταν καλό να μεταφέρετε ε, το ποσό αυτό, αντί να επιστρέφετε στο κράτος μέλος, στην επόμενη οικονομική χρήση, στην επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάλιτιτς. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς σας αναφέρω ότι είναι αναπόφευκτο αυτό το performance budgeting. Θα πρέπει να επιδιώκουμε κάποια αποτελέσματα. Θα πρέπει να βρίσκουμε κάποια μέτρα και κάποιους δείκτες για να βλέπουμε αν πετύχαμε πρόοδο, αν πετύχαμε αυτό το οποίο θέλαμε για κάθε πολιτική μας. Και επίσης συμφωνώ από αυτά που είπε ο μιλητής Uh, uh, πάρα πολλούς φραγμούς για την ορθή εκτέλεση του performance budgeting. Οπότε γι' αυτό ορίζουμε το, το, το πώς θα γίνει η μέτρηση, η αποτίμηση και αν κάτι είναι εύκολο και τίνουμε να το κάνουμε συχνά γιατί έχουμε αποτελέσματα, μα τότε αν έχουμε κάτι καινοτόμο, ε, τότε νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα. Για να ολοκληρώσουμε, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Μπολ. Τι, πώς σας εμπνέουν όλα αυτά που ακούσατε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα. Εμεί δεν τα χρησιμοποιούμε καθόλου στη Βάδη Βιτεμβέργη. Πραγματικά δεν υπάρχει κάποιο τομέα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν ε, σωστά. Αλλά πράγματι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ε, άλλα προβλήματα, ότι σε κάποιους τομείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη, όμως με τα έργα χρειάζεται κάποιες φορές να ε, καταθέσουμε μια τοποποίηση και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό έχει νόημα. Κατά τα λοιπά, πραγματικά μίλησα στην ψυχή μου, ε, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα ε, η καινοτομία χρειάζεται περισσότερο αέρα, αν θέλετε, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Συμφωνώ πολύ. Κύριε Γκρέσλε, έμαθα και εγώ κάτι για την καινοτομία. Θα πρέπει να τα κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά σε σχέση με τα άλλα τμήματα. Ε, δεν θέλω να στενοχωρήσω τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών. Έχουμε τις κατευθυντέ γράμμες, έχουμε το δημοσιονομικό κανονισμό, έχουμε το κανονισμό ε, για το ΕΚΤ και τα διαθωτικά, πάρα πολλά σελίδες, πάρα πολλές παράγραφοι. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά. Έχετε εσείς ε, διαβάσει τα σχετικά. Ναι, πράγματι, και ένας συνάδελφος ε, ε, που έκανε μια ομιλία στις Βρυξέλλες έφερε ένα, μια δεσμίδα 2.500 σελίδων έγγραφα και τα έβαλε πάνω στο τραπέζι για να καταλάβουμε την πολυπλοκότητα. Κύριε Γκρέσλε, πράγματι αυτό είναι το πρόβλημα Μόλις αυτούς τους κανόνες τόσοι πολλοί και διαφορετικοί κανόνες. Πραγματικά αυτό συνιστά ε, υπερβολικό φόρτο. Και νομίζω ότι και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ίσως και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ο Πρόεδρος. Είναι κομβικό το σημείο αυτό. Γιατί εδώ έχουμε δύο είδους επιδόσεις. Καταρχήν, είναι η κυβερνητική που θέλει τις ε, ποσότητες που έχουν καταθέσει στον προϋπολογισμό να τις παρυπήσει. Λοιπόν, έχουμε το πολιετές αυτό, όπου ο καθένας δανείζει, ουσιαστικά αυτό κάνει, και προσπαθεί να ε, πάρει τα χρήματά του πίσω. Έτσι, για να το πω πολύ απλά. Με συγχωρείτε δηλαδή που το λέω έτσι, αλλά αυτό συμβαίνει. Βάζουν χρήματα και περιμένουν να τα πάρουν πίσω. Το δεύτερο είναι δράσεις που έχουν κάποια χρησιμότητα, για την απασχόληση, για την κοινωνική συνοχή και για τη γενικότερη δυναμική της οικονομίας. Έχουμε λοιπόν φτάσει σε ένα επίπεδο όπου είναι τόσοι πολλοί οι κανόνες που εφαρμόζουμε τους κανόνες για κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή, εντάξει, όντως δημιουργεί αυτό θέση απασχόληση στις περιφερειακές διοικήσεις, στις τοπικές διοικήσεις, δημιουργεί απίστευτο εκνευρισμό και φαίνεται η Ευρώπη να είναι μια ε, αδυσόπιτη γραφειοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα και μπορούμε να περάσουμε τώρα στο ΣΕΠΣ για να μιλήσουμε για το ΕΦΣΙ. Σας δίνω το λόγο κύριε Νούνιες. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να μιλήσω στις επιτροπές σας. Τι έψη, τι εσύφ. Ε, σχεδόν ίδια είναι. Ένα γράμμα διαφέρει. Παρ' όλα αυτά όμως, παρ' όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό τα συζητούμε την κατάλληλη στιγμή. Διάβασα ένα βιβλίο επιστημής φαντασίας και μετά αποφάσισα ότι θα πρέπει τα πράγματα να τα βλέπουμε αποστασιοποιημένα. Όλοι εσεί εδώ είσαστε οι ειδικοί. Ε, μπορεί να καταλάβετε. Οπότε για αυτό και θέλω τώρα να δούμε το δάσος και όχι το κάθε δέντρο αυτού του μεγάλου δάσους των κανόνων. Να δούμε το ΕΦΣΙ και το ΕΣΥΦ. Ταμείο Στατικών Επενδύσεων και το Ταμείο ε, Διαρκτικής Πολιτικής και Επενδύσεων. Α, να, δουλεύει, δουλεύει. Για να δούμε τώρα με τις διαφάνειες. Πρώτα απ' όλα να δούμε τις βασικές αρχέ, Κάτι το οποίο πάντοτε είναι μια καλή ιδέα. Γιατί πάρα πολλά έχουν αλλάξει. Έχουμε μια διαδρομή 20 ετών που αλλάζουμε τον προϋπολογισμό, τον ε, τροποποιούμε, τον διορθώνουμε, τον προσαρμόζουμε, ε, προσπαθούμε να εξαντλήσουμε ε, τα, τα πλαφόν για να κάνουμε ακροβατικές προσπάθειες. Για πολλές φορές δεν ενεργούμε λογικά. Οπότε πολλές φορές αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου, αλλά δεν ωφέλουν και πολύ. Δεν αλλάζουν οι διαφάνειες. Α, μάλιστα. Είδατε, έχω θέμα με την τεχνολογία. Δεν είμαι τόσο καλός. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα αυτό του είδους την πολυπλοκότητα αυτόν τον γαλαξία που σας απελπίζει και βλέπετε εδώ τα περισσότερα ε, είναι εξωτερικά, είναι εκτός του προπολογισμού και βλέπουμε ότι έχουμε γαλαξία μέσα στον γαλαξία. Τη μία πολυπλοκότητα μέσα στην άλλη. Αν μου μια ματιά θα σας πιάσει απελπισία και θα πείτε και τι κάνουμε τώρα. Οπότε και τώρα έχουμε νέους κανόνε ή κανόνε που ρυθμίζουν τους άλλους κανόνες. Ε, εδώ πέρα, πήγε κάτι στραβά γιατί είδαμε ότι μπορέσαμε εδώ να κάνουμε κάποιους κανόνες που είναι εκτός των στόχων μας. Έχουμε αυτήν την πολιτική της συνοχής και την έχουμε διαιρέσει σε διαφορετικές κατηγορίες και έχουμε διαφορετικούς στόχους. Οπότε τώρα έχουμε διαφορετικούς κανόνες γιατί το σύστημα αυτό έχει πολλές διαφορετικές εφαρμογές και βλέπω ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των θεσμικών οργάνων και θα πρέπει κανείς να βγάλει ένα εργαλείο από κάθε στόχο. Όλα αυτά είναι πολύπλοκα. Επομένως ε, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες, διαφορετικοί πόροι για κάθε, κάθε στόχο, κάθε εργαλείο. Όχι δεν λέω ότι πρέπει να το στρατούς, αστυνομίες, νοσοκομεία, αλλά έχουμε κάποια εργαλεία τα οποία είναι χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Επομένως, εκμεταλλευόμαστε την προσθέμενη αξία γιατί προσπαθούμε να μοιράσουμε το καρβέλι μεταξύ όλων των σκοπών μας. Όμως από την άλλη μεριά, ακόμα και αν δεν μας αρέσει υλικά, τα γεγονότα προχωράνε. Επομένως, Έχουμε θυμότητα επίπεδου, εξετάζουμε την ευελιξία. Θα πρέπει να πω εδώ πέρα πλούστευση, αλλά θα ήταν πολύ μακροσκελές. Και αυξάνονται οι, οι ανάγκες μας και έχουμε και το Brexit. Όμως γλώσσα λανθάνουσα. Την αλήθεια λέει γιατί τελικά με το Brexit θα οδηγηθούμε σε πιο ισχυρό προϋπολογισμό. Και τι γίνεται τελικά, πάμε σε πιο είδου ευέλικτες παραχές, ενισχύσεις, ε, θολώνουν τα, όρια μεταξύ διαφορετικών τίτλων του προϋπολογισμού, κεφαλαίων, γιατί τα λέμε εδώ και χρόνια, όπως είπαμε, θα πρέπει να περισσότερη ευελιξία. Θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στη διάθεση των πόρων και όλα αυτά θα πρέπει να προσπολήσουν σοβαρά. Αλλά κινούμεθα σε μια συγκυρία κρίσης γιατί έχουμε όλα αυτά τα οποία τα, λέμε εδώ και τόσα χρόνια και ακόμα και αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ, ακόμα και εκεί πριν ε, δημιουργηθεί, δέκα χρόνια πριν υπήρχε η ιδέα και έχω δει τα σχετικά έγγραφα, εδώ λέγανε ότι χρειάζεται. τα ίδια για τον προπολογισμό. Θυμάμαι, είχε πέσει αυτή η ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο ε, ταμείο της χώρας. Οπότε τελικά λέμε ότι θα έχουν περισσότερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη κατανομή των πόρων και να ξαναγυρίσουμε πάλι στα βασικά θέματα για την απλούστευση. Θα πρέπει να απλουστεύσουμε, ούτως ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την πολυπλοκότητα και δεν χρειάζεται να έχουμε ε, με την απλούστευση περισσότερη πολυπλοκότητα. Άρα να απλουστεύσουμε ό,τι χρειάζεται και έτσι να διαχειριστούμε τα πιο μπερδεμένα, τα πιο δύσκολα και να έχουμε έτσι καλύτερα μέσα και εργαλεία για να διαχειριστούμε την πραγματικότητα. Οπότε για σκεφτείτε το λίγο. Είναι απλός ο κόσμος. Έχουμε αυτές τις επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις. Και αυτέ κινούνται από την πολιτική μας, από τα διάφορα ταμεία, κατόπιν έχουμε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, τα οποία παρά το ότι αποσκοπούν ε, σε κάποιους στόχους που έχουμε, είναι κάτι το πιο απαιτητικό, οπότε γι' αυτό το λόγο έχουμε δύο συστήματα. Αυτά τα δηλαδή εκατοντάδες έχουμε, αλλά ουσιαστικά αυτά είναι τα δύο βασικά. Δηλαδή σε αυτές, σε αυτές τις ε, ενισχύσεις ε, λέμε ότι καλύπτουμε τις ε, υποδομές, καλύπτουμε το capacity building, την υγειονική ανάπτυξη, την καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία στην αγορά, μετά, έχουμε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, τα οποία αφορούν τις υποδομές, την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την ε, καινοτομία. Είναι αυτά τα δύο μέσα, τα δύο εργαλεία που έχουμε. Α, είχα και μια εικόνα από κάτι ψαλίδια, που δεν, τη βλέπετε όμως. Αλλά κατά... Α, να τα, να τα, ψαλίδια. Το ψαλίδι, βλέπετε ότι με αυτό το ψαλίδι έχουμε ε, αυτού του είδους ε, τον έλεγχο και έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πάνε χαμένα τα λεφτά και ότι είναι θωρακισμένος ο προπολογισμό από τους κινδύνους, οπότε από τη μία μεριά έχουμε αυτή την εικόνα της περιφέρειας, της περιοχής, τους τομείς, του, ε, του, του, τους διάβλους της χρηματοδότησης που πάνε εκεί στις χώρες, στις περιφέρειες, στις, με διαφορετικούς κανόνες. Μετά έχουμε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, οπότε τελικά η λειτουργία είναι η ίδια και για τις ενισχύσεις για τις χρηματοδοτήσεις τα χρηματοοικονομικά. Αλλά όλα αυτά έχουν γραφειοκρατία και έχουμε όμως διαφορετικούς κανόνες για τον ίδιο σκοπό. Έχουμε τις ΜΜΕ, για το ΕΦΣΙ, έχουμε το ΕΦΣΙ για την καινοτομία, επομένως Τώρα έχουμε αυτή τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση και αναθεώρηση η οποία είναι πολύ μακριά, γαλαξίες μακριά. Είναι, το, το λέγαμε το, από το 10, είναι μια μεγάλη βελτίωση και έτσι μπορούμε να έχουμε δρόμο μπροστά μας το 2020 και λέω ότι βοηθά γιατί ξεπερνούμε έτσι πολλούς φραγμούς. Υπάρχουν πολλά θέματα που δεν τα συζητούμε γιατί εδώ προκύπτουν διάφορα θετικά. Έχουμε και τα καταπιστεύματα. Δεν τα ενέταξα εδώ στον κατάλογο, αλλά είναι τα trust funds, τα καταπιστεύματα σαν την ασπιρίνη. Γιατί έτσι ξεχνάει κανείς την ασθένεια από την οποία πάσχει. Γιατί πολλές φορές τα πλαφόνια δεν είναι ρεαλιστικά. Και με τα καταπιστεύματα αποφεύγει κανείς στην ουσία των προβλημάτων. Οπότε και έτσι πάνε στον κάθονα χρήστον οι αρχές μας για να τηρούμε τα προσχήματα. ας πούμε έχουμε αυτό το 1% που είναι τα Άγια των Αγίων και άλλα που δεν θέλουμε να θίξουμε. Οπότε παίρνουμε την ασπιρίνη που δεν είναι όμως ε, αποτελεσματικό φάρμακο. Τώρα βλέπουμε την ε, βελτίωση, η βελτίωση όσον αφορά τον δημιουργικό κανονισμό. Αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι η άριστη των λύσεων γιατί θα πρέπει να καταφέρουμε έτσι κάτι άλλο. Να, τώρα σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια θα δείτε. Έρχεται το Brexit, η συζήτηση για το ποιος πληρώνει. Ένα σωρό προκλήσεις. Και πάρα πολύ σωστά τα είπε ο των Διευθυντής για τον προϋπολογισμό σε κάποια συνάντηση πρόσφατα. Είναι δισεκατομμύρια. Ποιος θα πληρώσει, ποιος θα επιστρέψει τα χρήματα. Μα και ακόμα και έχουμε 50 50 ε, δις, εγώ νομίζω ότι θα αξίζει τον κόπο. Γιατί δεν πειράζει. Γιατί ανησυχείται Ο προπολογισμό παραμένει πάρα πολύ πλούσιος. Ε, πρόκειται για θέματα και μας βοηθά να βρούμε λύσεις και να μας πιάνει ο πανικός. Επομένως, χρειάζεται καλύτερη χρήση των παροχών σε διαφορετικούς τομείς, ευθυγράμμιση των κανόνων, να μην ε, Έχουμε προβλήματα με το τι, γίνεται με την ανάπτυξη της υπαίθρου, πρόκειται για, για χωριό ή όχι. Είναι, είναι ένας δρόμος που θέλουν να φτιάξουν για το χωριό. Πού να πάει κανένας στην περιφερειακή ανάπτυξη, στη γεωργία. Τι ε, διαδικασίες χρειάζονται. Άρα χρειάζεται εναρμόνιση, ευθυγράμμιση κανόνων. Επίσης θα πρέπει να γίνει κατανομή των πόρων επί τη βάση των αναγκών και της ποιότητας των προγραμμάτων. Ε, εδώ έχουμε κάνει βήματα πρόοδου που είναι θετικό. Κάποια, κάποια βήματα πρόοδου. Αλλά θα πρέπει να μειωθεί η πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών ε, εργαλείων. Θα πρέπει να ε, είναι το βασικό κριτήριο η ζήτηση όσον αφορά τη χρήση της χρηματοδότησης γιατί αυτό μας περιορίζει και το κόστος. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά από ότι τις ενισχύσεις της παροχής εν προκειμένου. Και θυμάμαι ότι υπήρχε μια χρηματοδότηση που αφού εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και από άλλα όργανα, αλλά μπήκαν τόσοι πολλοί περιορισμοί στη χρήση αυτών των πόρων που τελικά κανένας δεν θέλησε να γίνει επιλέξιμος. Επομένως, ε, θα πρέπει να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το κόστος και τελικά έχουμε ε, ένα καλάθι, οπότε ε, έχουμε ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο και να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένους ε, κανόνες, προσθετικότητα, ένα κλάδο και επίσης να δούμε πώς θα φροντίσουμε και τις ΜΜΕ και την, τις υποδομές. Να μην έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές διαδικασίες, αυτό ακούγεται σαν ένα όραμα, θα πάρει χρόνο. Ξέρω ότι ζητάω πολλά, αλλά τουλάχιστον το, το, σκέφτομαι. Να, ποιο είναι το όνειρό μου. Απλουστευμένο προπολογισμό, έχουμε τι ενισχύσει, ε, ανθρώπινοι πόροι, υποδομέ και από την άλλη μεριά έχουμε τα, τα μέσα, τα χρηματοοικονομικά και έχουμε επίση και αυτό το παράθυρο τη ανάπτυξη. Γιατί το λέω έτσι. Μπορούσαμε να το πούμε και αλλιώ, γιατί φτιάξαμε το ΕΦΣΙ και λέει ο κόσμο ότι το εύση δεν πρόκειται να καλύψει τις ε, δυσκολίες των περιφερειών. Μα το ΕΦΣΥ δεν αποσκοπεί σε αυτό. Εάν θέλετε να καταφέρετε κάτι τέτοιο θα πρέπει να φτιάξετε ε, κάτι άλλο. Το αντιμετωπίζει τους κινδύνους αυτών των περιοχών. Ε, άρα το κριτήριο είπαμε ότι είναι η ζήτηση. θα πρέπει κανείς επίσης να ελκύσει επενδυτές να μην χάσει κανείς την αξιολόγηση του 3α, τότε θα τα πράγματα χειρότερα. Και επίσης να δούμε τι γίνεται, τι κάνουμε στη μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι εκτός αυτής. Άρα για τις υποδομές ε, έχουμε κάποια όργανα και, να έχουμε κοινού κανόνες να τα συνδυάσουμε αυτά και αν είναι απλουστευμένος ο προϋπολογισμός και οι διαδικασίες, τότε οι περιπλοκότητες αντιμετωπίζονται. Και ο έλεγχο γίνεται ευκολότερο. και βάζω τελεία. on aura un Άρα θα έχουμε κανονισμό 10 σελίδων ή και λιγότερο. Μα αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Ξεκίνησε η Επανάσταση. Κυρία Γκρέσλε. σκέφτηκα μήπως πρέπει να παραιτηθώ, τέλος πάντων. Πώς να το πω. Έχετε απόλυτα δίκιο με την περιγραφή της κατάστασης όπως την κάνετε. Και το πρόβλημα είναι ότι όλα είναι δυνατά και τα αντίθετά τους ταυτόχρονα. Και αν προχωρήσουμε έτσι, και αν αντί να τα στεγανοποιήσουμε και να τα ξεκαθαρίσουμε, τα μπερδεύουμε τα πράγματα, δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από αυτή την κατάσταση. Μετά από 13 χρόνια, ε, αν έχουμε, διαπιστώνω χιλιάδες εξαιρέσεις για ένα κανόνα, Δυσκολεύουμε τα πράγματα, δεν υπάρχει ορατότητα ε, για τους ε, δικαιούχους, για τους αγωδεξιούς. Έχουμε έξι γενικές διευθύνσεις που επεξεργάζονται τα αναπτυξιακά κονδυλέξη, διαφορετικές βασικές πράξεις, κατευθυντήριες γραμμές, ε, διαδικασίες, έντυπα και το καθεξής. Όταν λοιπόν οι δικαιούχοι έχουν δύο-τρία σκορβανάδες αν θέλετε από τους οποίους να αντλήσουν χρήματα και έχουν 5-6 ανθρώπους ε, που πρέπει να ασχολούνται μόνο με τους κανόνες και τις αλλαγές των κανόνων και με το single book ε, μπορεί να μην λύνονται όλα τα προβλήματα, αλλά τέλο κάτι, κάτι γίνεται. Πρέπει να υπάρξει ε, μια συγκέντρωση των πραγμάτων. Εγώ συμφωνώ, για, σας ευχαριστώ για αυτό το άκρος πολύπλοκο γράφημα, το πάρα πολύ εύγλωτο Το θέμα είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε ε, την ε, ε, δυνατότητα να έχουμε ευέλιξη με τον υπολογισμό. Ε, ίσως και στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Κάναμε ήδη κάποιες προσπάθειες, πρέπει να δούμε τι μπορούμε ακόμη να κάνουμε πιο απλό. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δική σας δουλειά. Μα ξέρετε αυτό το πίνακα, αυτό το γράφημα το έχει φτιάξει η Επιτροπή Προϋπολογισμού, ξέρετε. Ε, όχι, ο... ο κύριος Φερνάνδης, σας ευχαριστώ πολύ. Να σας πω πως το πίνακα αυτό το χρησιμοποιούμε ως η απόδειξη πως ακολουθούμε την οδό της επιπλοκής. Και κάθε φορά πολλαπλασιάζουμε περίπλοκες διατάξεις και εμείς ως εισηγητές θα πρέπει τελικά να κάνουμε την αντίστροφη διαδρομή και να ξεκινήσουμε να απλουστεύουμε. Και ίσως δεν θα είναι υπερβολικά δύσκολο. Υπάρχει κάτι ακόμα. Για μιλά, ε, μιλάμε εδώ για δικαιούχους και τα λοιπά. Θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτήν την περίπλοκη κατάσταση και την περίπλοκη, τις παρέπλοκες διατάξεις που ακολουθούν σε επίπεδο εθνικών διατάξεων που περιπλέκουν ακόμα περισσότερο και μετά ακολουθούν η περιφερειακή νομοθεσία που περιπλέκει και ακόμα περισσότερο. Και τελικά οι βασικοί μας στόχοι δεν επιτυγχάνονται. Υπάρχει κάτι ακόμα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να με συγχωρέσει, αλλά με συγχωρείτε. Αυτό το τόσο περίπλοκο δεν κατάφερε να λύσει το τεράστιο πρόβλημα που είχαμε με τις πληρωμές. Γιατί το 2014 είχαμε 23 δις ε, πληρωμών που δεν είχαν πληρωθεί. Φανταστείτε λοιπόν αν μπορούσαμε να τρέξουμε τον κανονισμό μας με καλούς ρυθμούς. Δεν είχαμε χρήματα για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και νομίζω ότι η κακή εκτέλεση βοήθησε με πραγματικά βαθύ τρόπο να βελτιώσουμε την κατάσταση με τις πληρωμές. Δηλαδή μιλάτε για τον ε, κανονισμό ο οποίος οδηγεί σε κάποια αυτορύθμιση της χρήσης του προϋπολογισμού. Ναι, λέει ο κ. Φερνάντες. Ακόμα και στο γαλαξία έχουμε τις επιδοτήσεις και από την άλλη είναι ένα άλλο γαλαξία που είναι η, ε, τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μην ξεχνάτε και το γαλαξία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολλά εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν και στα διαφορετικά ταμεία έχουμε και την καλή δυνατότητα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα επενδυτικά εργαλεία και μηχανισμούς που δεν είναι περίπλοκο γιατί αν κοιτάξει κανεί το ολόκληρο σχέδιο θα πει ότι είναι υπερβολικά πολύ σύνθετο, αλλά αν κάνει focus θα δει πως αυτό ουσιαστικά περιορίζει το πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Είναι όμως αλήθεια πως θα έπρεπε για να μεγιστοποιήσουμε να απλουστεύσουμε. Έτσι ώστε να έχουμε τη μέγιστη απόδοση του κάθε ευρώ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον ορισμό για την προσθέμενη αξία, αλλά αυτή ακριβώς είναι η προστιθέμενη ε, αξία, αλλά μην με αντιγράψετε, σας παρακαλώ πολύ. Αυτός είναι ο δικός μου ορισμός. Και θα ήθελα να πείτε ποιος είναι ο δικός σας ορισμός και αν υπάρχει κάποιος ορισμός της προστιθέμενης αξίας. Και αν υπάρχει, ρωτώ το εξής. Αυτό το τελευταίο και Grants and Financial Instruments, αυτό συνδυάζεται με τις επιδοτήσεις που έχουμε και για το πολιετές πρόγραμμα. Θα μπορούσαμε αυτά να τα προσθέσουμε ως υποδομές, ανθρώπινο κεφάλαιο, κοινωνικά κτλ. Και μην ξεχνάμε και τη γεωργία βέβαια. Μήπως έτσι λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε το πολιετές πλαίσιο. Δεν έχω τίποτα. Ε, και βέβαια μπορούμε να ακολουθήσουμε με το είδος πρόσθεσης που κάνουμε σήμερα. Έχει λειτουργήσει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η πρόταση αυτή θα έχει κάποιες επιπτώσεις για το format που, το format που χρησιμοποιούμε για τις πολιτικές ε, προοπτικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, η κυρία Μάλετη, επόμενη ομιλήτρια. Θα ήθελα να τονίσω, το όταν μιλάμε για απλούστευση και αλλαγές στον προϋπολογισμό, θα έπρεπε πάντα να έχουμε κατά νου πως από τον προϋπολογισμό χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το βασικό ερώτημα που είναι τι, που και πώς χρηματοδοτείται. Και αν θέλουμε να δούμε τι χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό, τότε χρειαζόμαστε ταξινόμηση των προγραμμάτων, δηλαδή προγραμματική και πολιτική προσέγγιση, ε, ε, αναπρότζεκτ προσέγγιση και το τι χρηματοδοτείται σε οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή ε, κεφάλαια, υλικά, εξοπλισμοί, ε, υποδομές, για παράδειγμα. Επίσης, και μια τοπική ταξινόμηση και πώς αυτό το πώς χρηματοδοτείται έχει να κάνει με την πηγή χρηματοδότησης. Δηλαδή ποια μέσα, αν είναι χρηματοδοτικά εργαλεία, αν είναι επιδοτήσεις, ενισχύσεις, άλλου είδους πηγές. Άρα λοιπόν τα έγγραφα θα πρέπει να είναι απλά οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι απλές, αλλά θα πρέπει να απαντούν αυτές τις βασικές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. και Ζήστε, το λόγο. Νομίζω ότι ένα από τα συμπεράσματα το... της συνα... σημερινής συνάντησης είναι οι επιπτώσεις του κειμένου αυτού. Πόσοι θα το διαβάσουν αυτό το κείμενο. Πόσα μέλη του Κοινοβουλίου θα το καταλάβουν, ακόμα και από τη δική μας Επιτροπή, αυτόν τον κανονισμό. Ποιοι θα τον καταλάβουν και ποιοι θα τον διαβάσουν. Η κυρία Γκρέσλερ μέχρι σήμερα, ίσως και κάποιοι ακόμα. Όσο λοιπόν για τις επιπτώσεις, ο εισηγητής ήταν όπως πάντα πολύ σαφής, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε και το γνωρίζουμε και είναι κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και χρόνια, είναι Κάτι το οποίο κανείς δεν αρνείται και κανείς δεν θέλει να αλλάξει. Για ποιο λόγο, υπερπείου η απλούστευση, ποιο ωφελείται από την απλούστευση, για χάρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή για τους δικαιούχους. Μπορούμε να φανταστούμε πως ω επίπτωση του, του, της ρύθμισης αυτής να έχουμε μια εργαλειοθήκη που θα επιτρέπει σε κάποιον που θέλει κάτι να κάνει να πάει κάπου και να πει θέλω να κάνω το χ. Πώς μπορείτε να το χρηματοδοτήσετε. Πού είναι η εργαλειοθήκη, ποια είναι η περίσταση, τούτο το ταμείο, το άλλο. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε το τι κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παντού. Όχι, ένα απλό ε, σύστημα, μία πολύ απλή εργαλειοθήκη, διαφορετικά όλα τα υπόλοιπα είναι άχρηστα. Και δύο σχόλια, το λέω και θα κλείσω. Πρώτα απ' όλα τώρα, δημιουργούμε μια ακόμα πιο περίπλοκη κατάσταση από ό,τι σήμερα. Δηλαδή, το να ε, μοιράσουμε έτσι την, την πολιτική συνοχή είναι απλώς το πρώτο βήμα. Γιατί τώρα προσπαθούμε, μετά το 2020, προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη διέρεση στην πολιτική συνοχή. Αυτό είναι. Και τώρα προσπαθούμε να δούμε ποιε γενικέ διευθύνσει θα κάνουν. Τι και ποιο επίτροπο θα κάνει τι. Και αυτό είναι σημερινό. Δεν είναι παλιό. Και το τελευταίο, Δυστυχώς Η ασπιρίνη είναι το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον προπολογισμό. Δημιουργούμε καταπιστεύματα, αλλά αυτά βρίσκονται εκτό προπολογισμού και δεν λύνουν το πρόβλημα. Αν, επειδή δεν μπορούμε να το εντάξουμε στον προπολογισμό, το βάζουμε σε ένα καταπίστευμα. Η ερώτηση είναι εξή. Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε αυτά που είναι σε καταπιστεύματα στον προπολογισμό και να απλουστεύσουμε, όχι το αντίστροφο. Συνοψίζω λοιπόν. Πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Πρέπει ο κανονισμός αυτός να είναι πολύ απλός για τον τελικό δικαιούχο να είναι όσο το πιο δυνατόν απλός και μια απλή εργαλειοθήκη. Τι μπορεί να χρηματοδοτήσει πιο project. Όπω είχε πει και ο Πρόεδρό μα, οι πολίτε ποτέ δεν θα καταλάβουν τίποτα και δεν θα παίρνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια αν είναι υπερβολικά περίπλοκε οι διαδικασίε για να τα ε, λάβουν. De comprendre Άντε να προσπαθήσει να καταλάβει τα οργανογράμματα των γενικών διευθύνσεων. Α πούμε, κάποιε γενικέ διευθύνσει τη Κομισιόν. Δεν καταλαβαίνετε βλέποντάς τα ότι και εμείς έχουμε αναγκαστικά πολύπλοκες διαδικασίες εξ αυτού. Μήπως θα έπρεπε κάποια στιγμή να ασχοληθούμε από κοινού και να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα, γιατί αυτή η πολυπλοκότητα ουσιαστικά καθρεφτίζει και τη διαδικαστική πολυπλοκότητα, την πολυπλοκότητα του δημοσιονομικού κανόνα, που είναι αποτέλεσμα της πολύπλοκης οργάνωσης κομισιών. Πάντως ήταν πολλά υποσχόμενη η παρέμβαση δεν ξέρω αν ε, ο εισηγητής θέλει να πάρει ξανά το λόγο, ίσως για μια σύσταση. Επαγόρευση να ναι, το πάρα πολύ γρήγορα, όπως βλέπετε. Μπορείτε να συζητείτε τους τίτλους, ε, τις ε, κατηγορίες, δική σας είναι η απόφαση. Αλλά Υπάρχει πραγματικά μεγάλη πλειοποκότητα, πολλά προβλήματα που μας επηρεάζουν ναι. και σε συναντήσεις που έχω για την ευφύ τεχνολογία βλέπω ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν ε, ασχολείται με το δίκτυο παροχής ενέργειας η DG Energy αλλά DGI, είτε ICT ή κάτι, κάποια άλλη παρότι μπορεί να είναι αστικό σχέδιο. Και σε ό,τι αφορά τη μοναποθετική θηρίδα για τους ε, δικαιούχους, ε, τους στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα. Επειδή ασχολούμαι όμως με τις πόλεις τώρα, καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Χρειάζεται μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε τα διάφορα μπλοκ για να δούμε αυτή την ε, πολυπλοκότητα, πώς θα την αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι ολοκληρωμένη, ενοποιημένη πολυπλοκότητα, integrated complexity. Και αυτό είναι το τελευταίο μήνα. Αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ. Πάντως σίγουρα μας εμπνεύσατε. Ε, για να δούμε τι γίνεται με τα, την ιστορική κουζίνα εδώ στις Βρυξέλλες να καλωσορίσω τον επόμενο ομιλητή σε σχέση με το θέμα ε, Service Level Agreement και την εξωτερική ανάθεση θα μας μιλήσετε. Κύριος Μονάτ, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ που δίνετε δυνατό στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των διαφόρων οργανισμών. Ε, να είναι εδώ για να σας παρουσιάσει κάποια πράγματα. Εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω αυτό το θέμα της εξωτερικής ανάδυσης καθήκων της τοπίσει και να το βάλω στο πλαίσιο. Ξέρετε ότι οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη. Μ' ακούτε? Okay. Uh, strategy and the Juncker Commission agenda για τη στρατηγική 2020 και τη θεματολόγιο Juncker. Και στόχος βέβαια είναι να ε, ωφελήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Για να τις πετύχουμε, έχουμε ήδη αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Στο πλαίσιο της εντολής μας ε, υπάρχει συνεργασία, συντονισμός, ε, συνένωση πόρων, τεχνικών, αλλά και πυργνωμοσύνης και συνεργασία με εθνικές αρχές, βιομηχανία κτλ. Άρα ήδη κάνουμε αυτή την εξωτερική ανάθεση καθηκόντων και δραστηριοτήτων. Επομένως, μπορεί να κεφαλαιοποιήσει η Ένωση ε, στην ε, αξία των οργανισμών αυτών και για την επίτευξη των στόχων, των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο ωφέλη τελικά για τους πολίτες. Και έχουμε και αυτό το δίκτυο που σας περιέγραψα, μέσω του οποίου συνεργαζόμαστε. Το σχέδιο ε, τη εκθέση απαλλαγή για το 2015 σε σχέση με του κλειστικού οργανισμού ήδη σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι οργανισμοί αυτοί με βάση θεματικέ ομάδε ήδη συνεργάζονται, καλούνται βέβαια να συνεργαστούν πιο στενά στο πλαίσιο τη θεματική ομάδα για συνέργειε ε, αλλά και για συνεργασία στους κοινούς τομείς πολιτική. Βασική αποστολή και στόχοι είναι πέντε θεματικές ομάδες. Πρώτο, ασφάλεια και άμυνα. Το χώρος ελευθερίας δικαιοσύνη ασφάλειας. Ευημερία πολιτών. Στήριξη καινοτομίας και επιχειρήσεων της Ένωσης και εποπτεία χρηματοπιστικών συστημάτων. Αυτές είναι οι ομάδες. Και ξέρετε ότι έχουμε 44 αποκεντρωμένους οργανισμούς και κοινοπραξίες. Έχουμε προβλησμένο ακόμα 2 δις που είναι κάτω από το 0,8% του συνολικού ετήσιου προπολογισμού της Ένωσης. Και έχουμε γύρω στα 5.500 άτομα προσωπικό το 2016. Θέλουμε λοιπόν την βελτιστοποίηση και των, πόρων και την ε, περισσότερη εξωτερική ανάθεση. Έχουμε το άρθρο 57 στην πρόταση της Κομισιόν, η οποία βάζει νομική βάση για την εξωτερική ανάθεση. Επιτρέπει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των οργανισμών μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Shared το λέμε εμείς αυτό. Η συμφωνία ε, αυτή στο άρθρο 57 λέει ότι το Service Level Agreement θα πρέπει να βοηθά την υλοποίηση του προπολογισμού, ιδίως όταν αυτά τις διοικητικές ε, πιστώσεις, παροχή προϊόντων, εκτέλεση έργων, εφαρμογή κτηριακών συμβάσεων. Επίσης αναφέρεται ότι με τη συμφωνία αυτή θα ανακτάτε το κόστος του κύριων του έργου. Και υπάρχει και ο μηχανισμός που βασίζεται στην αρχή της μία αποκόμισης ωφέλους για την ανάκτηση του κόστους αυτού. Στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, αυτός ο επιμερισμός ε, είναι κλειδί αν θέλουμε βελτιστοποίηση πόρων, ανθρώπινων και υλικών. Έχουμε τον χρηματοδοτικό, ε, μάλλον τον δημοσιονομικό κανονισμό, που δεν προβλέπει ρητό αυτό τον επιμερισμό ή τέλο πάντων τη συνένωση πόρων εκτό από εξωτερικού ελεγκτέ ή κοινοπραξη, ή μάλλον κοινή διοργάνωση διαγωνισμών μεταξύ των οργανισμών. Αλλά περιορισμένο το εύρο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ε, σε δώσουν περισσότερες υπηρεσίες για την πληροφορική, για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, για τις προσλήψεις, για τους ανθρώπινους πόρους, καθώς και για κάποια επιχειρησιακά καθήκοντα. Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν γιατί δίνει τη δυνατότητα στις ε, υπηρεσίες και οργανισμούς να έχουν πιο αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Όμως, με βάση την πρόταση της Κομισιόν, μόνο για οριζόντιες υπηρεσίες ή διοικητικέ υπηρεσίες προβλέπεται αυτός ο επιμερισμός. Εμείς θα θέλαμε να επεκταθεί και σε άλλες υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση να μην περιοριζόμαστε στους διοικητικούς, ε, στα διοικητικά καθήκοντα. Η εκτέλεση του Παπαλισμού θα μπορούσε να εκχωρηθεί από τον ε, εκτελεστικό διευθυντή ενός οργανισμού σε έναν άλλο. Είναι και αυτό μία επιλογή που μπορούμε να μελετήσουμε. Για τη σύναψη της συμφωνία τώρα. Αν συναυθεί αυτή η συμφωνία θα έχουμε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, θα έχουμε εξοικονόμηση πόρων, συνέργειες. Αυτό είναι πολύ σημαντικός στόχος. Δεν είναι μόνο η ανάκτηση του κόστους. Και επειδή όλο και μεγαλύτερο είναι ο φόρτο εργασίας και λιγότερο του προσωπικού, απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία στους ε, οργανισμούς για να μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των πόρων. Η εξωτερική ανάθεση μόνο όταν θεωρείται, το outsourcing δηλαδή, θεωρείται μόνο, επιτρεπτό μόνο όταν είναι απόλυτα απαραίτητο με τον ε, ε, ισχύοντα δημοσιονομικό οργανισμό, θα έπρεπε να αλλάξει αυτή η διάταξη, πιστεύουμε. Γιατί και οι εξωτερικοί ανάδοχοι ουσιαστικά του ίδιου στόχου ε, επιδιώκουν. Βέβαια δεν είναι όλοι επιτυχημένοι. Πολλέ φορές έχει αφιεστηθεί από το ελεκτικό συνέδριο η ε, αποτελεσματικότητα της ξέρχης ανάθεσης. Γιατί απεδείχθηκε ότι αυξήθηκε το κόστος των οργανισμών. Άρα ανησυχούν οι οργανισμοί. Και με τροπολογία 59 πρόταση κανονισμού, άρθρο 69, συγγνώμη. σε ό,τι αφορά τι διατάξει της κανονικότητας και της νομιμότητας. Υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των τριών θέσεων οργάνων του 2012 σε ό,τι αφορά την εξωτερική ανάθεση του λογιστικού ελέγχου. Η ΕΚΑ είναι αρμόδια. Το Ευρωπαϊκό δηλαδή Ελεκτικό Συνέδριο. Τρόπο 69 λέει ότι όλες οι πτυχές εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου και τα πορίσματα πρέπει να αποτελούν πλήρη, ε, να είναι υπό την πλήρη αποκλειστική ευθύνη του ελεκτικού συνεδρίου. Το ελεκτικό συνέδριο, επομένως, θα πρέπει να κάνει και τους διαγωνισμούς και να χρηματοδοτεί αυτούς τους εξωτερικούς ελέγχους βελτιστοποίηση πόρων έχει να κάνει και με τα έσοδα. Πολλοί οργανισμοί θα ήθελαν να κάνουν δραστηριότητα συνεργασία με άλλους φορείς της Ένωσης. Για παράδειγμα, ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με την Κομισιόν ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Άρα θα πρέπει να μπορούν να είναι οργανισμοί αυτοί δικαιούχοι για να μπορούν να έχουν αυτή τη συνεργασία. Μπορεί και να μην προβλέπεται στο καταστατικό ρητός, αλλά θα πρέπει να επιτραπεί. Μόνο αν υπάρξει ειδική παρέκκληση είναι εφικτό αυτό σήμερα και η οποία πρέπει να συζητηθεί με την Κομισιόν. Η απλούστευση και η ευελιξία είναι άλλοι στόχοι. Έχουμε πολύπλοκε δυσανάλυσε διαδικασίε. Δεν συμβεί στο προστιθέμενη άξια. Αυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν δημοσιονομική διαδικασία, για παράδειγμα, που χρειάζεται απλούστευση. Κατάργηση εσωτερικών ε, εσόδων ε, για ειδικό προορισμό. Το προβλέπει ή το προτείνει τέλο πάντων το ελεγκτικό συνέδριο. Θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πραγματική ε, προσέγγιση ανάλυσης κινδύνων εξάντε. Με τον δημοσιονομικό κανονισμό προβλέπεται σήμερα άμεσο σύστημα χρέωσης. Αλλά θα πρέπει για το ενίκιο, τα τηλέφωνα, το ρεύμα να ισχύει το ίδιο. Και όχι για το συγκεκριμένο είδος δαπανών που προβλέπεται μέχρι τώρα. Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού πραγματικά αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για ένα πιο σύγχρονο κόνσεπτ απλοί κανόνες που θα προσφέρουν ευελιξία. Και οι εκτελεστικοί διευθυντές βέβαια πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να αξιολογούνται βάσει των επιδόσεών τους, με βάση τους στόχους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Κύριε Μονάρ, σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω κάποιον το λόγο για ερώτηση προς τον κύριο Μονάρα. Άρα να συνεχίσουμε όπως προβλέπετε από το πρόγραμμά μας. Θέλει κάποιος το λόγο. Όχι. Επομένως, καλώς όρισε ο επόμενος ομιλητής μας. Ο οποίος θα μας μιλήσει για την εμπλοκή των πολιτών. Από πλευράς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Δημοσίας Δικήσεως του Μάστριχ είναι ο δόκτωρ Έντουαρντ Μπέστ. Σας ευχαριστώ πολύ είναι για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας για ένα θέμα το οποίο προσφέρει αρκετές προκλήσεις και για ένα κείμενο το οποίο έχει προταθεί για το οποίο, αν έχω καταλάβει καλά, ακόμα δεν έχετε καταθέσει τροπολογίες και ελπίζω πως ίσως να μπορέσω να πω κι εγώ κάτι χρήσιμο. Υπό την πίεση χρόνου που έχουμε θα ε, κατά κάτι την πρότασή μας και να σας πω ότι για κάποιους ίσως προξενεί έκπληξη το ότι σε κάποιο κανονισμό αναφερόμαστε στην εμπλοκή των πολιτών στη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά όταν ο στόχος είναι απλούστευση. Για άλλους τέτοιου είδους διατυπώσεις μπορεί να μοιάζουν απογοητευτικά ασαφείς ή μη δεσμευτικέ. Δηλαδή, δύναται να διαβουλευτούμε με τους πολίτες για... Ξέρετε πως σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει συνένεση πως η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην δημόσια πολιτική είναι ευκταία. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει συνένωση ότι συνένεση πως πρέπει να κάνουμε περισσότερα έτσι ώστε να προσεγγίσουν οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε δυνατό τρόπο. Είναι λοιπόν φυσικό και αξιέπαινο να προσπαθούμε να ενισχύσουμε την εμπλοκή των πολιτών στην εκτέλεση, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ε, προπολογισμού. Όμως, προσδοκίες και υποψίες θα έλεγα στο τρέχον πλαίσιο μαζί με τον εκνευρισμό για κάποιες άλλες πρόσφατες τέτοιου είδους προσπάθειες που έγινε η συμμετοχή πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σημαίνουν ότι ίσως θα έπρεπε οι φιλοδοξίες μας να μετριαστούν από την ε, προσοχή με την οποία πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα, έτσι ώστε αυτό το οποίο θα υποσχεθούμε μετά να, γίνει, να λάβει σάρκα και οστά. Οι κοινέ προσπάθειε θα έπρεπε να γίνουν έτσι ώστε οι πρωτοβουλίε για τη συμμετοχή των πολιτών θα είναι ε, και λογικές και θα τις διαχειριστούμε σωστά και πραγματικές και υπάρχει μια πλειάδα τρόπων με τον οποίο μπορεί να εξασφαλίσουμε αυτή τη συμμετοχή των πολιτών. Και επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι του προπολογισμού εφαρμόζεται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, δεν θα ήταν ενδεδειγμένο να συμπεριλάβουμε οτιδήποτε που να μοιάζει με νομική δέσμευση που να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ της τροποποίησης του κειμένου να γίνει ίσως λίγο πιο ενθαρρυντικό Δηλαδή, να πούμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τα κράτη-μέλη και οι οντότητες που εφαρμόζουν τον προϋπολογισμό ενθαρρύνονται να προωθήσουν όπου δει την εμπλοκή των πολιτών. Για την διατύπωση εδώ, νομίζω ότι ίσως είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί στο βαθμό που αναλαμβάνουμε δέσμευση και διατυπώνουμε υποχρεώσεις. Το πιο σημαντικό ενδεχομένως είναι να στηρίξουμε ε, πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν αυτή την ε, συμμετοχή και τη σωστή διαχείριση επιτόπου. Τι σημαίνει επιτόπου, σε τοπικό επίπεδο. Ναι, όντως. Έχουμε διάφορες εμπειρίες που λαμβάνουν χώρο σε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης και που έχουν καταγραφεί γιατί είχαμε μια επιτυχή ε, προσπάθεια συμμετοχή στην εκτέλεση του προπολογισμού. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το πώ κατανέμονται οι επιχορηγήσει για project σε ένα μάλλον ε, μικρό ε, εθνικό περιφερειακό επίπεδο και έχουμε κάποιες εθνικές εμπειρίες, Ιταλία, Γαλλία, Ενωμένο Βασίλειο, όπου έγινα να με τους πολίτες, για παράδειγμα για την αξιολόγηση των δαπανών. Και στην Ινδία, στην Ινδία ε, στην Ινδία έχουν αναφερθεί σε ό,τι κάνουμε, το MyGov εκεί ας πούμε λειτουργεί σωστά. Έχουμε λοιπόν αυτό τον, ε, όσους προωθούν τον ακτιβισμό των πολιτών που είναι σίγουροι πως τελικά θα προχωρήσουν τα πράγματα, θα γίνουν όλοι σε τοπικό επίπεδο και θα πρέπει να τα δούμε όλα υπό αυτό το πρίσμα. Θα μπορούσα εδώ να προσθέσω και κάποιες σκέψεις για τη διατύπωση της πρότασης που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη δημιουργία ενός υποβοηθητικού πολυεπίπεδου πλαισίου που θα βοηθούσε αυτή την πραγματική συμμετοχή επιτόπου. Να σας πω καταρχήν πως για την πιθανότητα επιτυχίας, να δούμε τα θετικά, προτείνω την παράγραφο που λέει πως θα διαβουλευτούν συζητούμε με τους πολίτες. Οι συγκριτικές μελέτες από την Ευρώπη και από τον υπόλοιπο κόσμο αποδεικνύουν πως η συμμετοχή και η εμπλοκή δεν έχει να κάνει με τη μία και μοναδική φορά που θα ε, μαζέψουν υπογραφές οι πολίτες ή θα γνωμοδοτήσουν. Το ζήτημα είναι όχι πώς θα ε, συλλέξουμε αυτές τις υπογραφές και θα τις ενοποιήσουμε, αλλά πώς μπορούμε αυτό να το εντάξουμε στις μακροπρόθεσμες διαδικασίες προβληματισμού, διαβούλευσης και λογοδοσίας που αποτελούν μια πιο ε, βαθιά έννοια εμπλοκή. Και μην ξεχνάμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν και στο τοπικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν καταγραφεί σε αρκετέ μελέτε για τον τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά ταμεία έχουν χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένα προγράμματα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Λόμπινγκ, για παράδειγμα, ε, χειραγώγηση. Στις προτινόμενες αλλαγές δίνεται η ενδεδειγμένη ε, σημασία στο να εξασφαλίζουμε τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των τοπικών ομάδων δράσης. Άλλος κίνδυνος σε όλα τα επίπεδα είναι χαμηλή συμμετοχή. Και το να επενδύει κανείς σε αυτές τις πρωτοβουλίες μπορεί τελικά να αποτύχει και να μην επιτύχει την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και λογοδοσία που επιδιώκονται. Και τελικά, αν δεν πάρουν την τροπή που θα επιθυμούσαμε τα πράγματα, ενδεχομένως θα υπάρξει και η απόρριψη, θεωρώντας πως αποτελεί απλώς ένα πολιτικό φτιασίδωμα, γιατί δεν οδηγεί σε ανάληψη υποχρεώσεων μεσοπρόθεσμα. Paragraph can be seen from different perspectives. Θα μπορούσαμε λοιπόν αυτή την παράγωγη να τη δούμε από διαφορετικέ οπτικέ γωνίε και το λέω αυτό συμπερασματικά. Υπάρχει ο κίνδυνο να μην δημιουργηθούν οι κατάλληλε προσδοκίε οι οποίε τελικά θα οδηγήσουν σε περισσότερο εκνευρισμό. Σω κάποια επαναδιατύπωση θα μπορούσε να γίνει, έτσι ώστε να έχουμε μια νέα προσέγγιση, ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο που θα εστιάζει σε αυτά τα οποία πραγματικά έχουν σημασία σε τοπικό επίπεδο. Διαβούλευση παρόλες τις αυξανόμενες προσπάθειες που κάνει στο πακέτο για την καλύτερη νομοθέτηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μια σειρά προγραμμάτων, τελικά αυτό θα γίνει κυρίως σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και δεν θα είναι μόνο θέμα μεμονωμένων πολιτών πώς μπορούμε να κάνουμε τη διασύνδεση με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να πετύχουμε τους άλλους στόχους που είναι τη συμμετοχική κατάρτιση προϋπολογισμού, δηλαδή μεγαλύτερη ταυτοποίηση ε, με το ευρωπαϊκό πλέγμα. Νομίζω ότι αυτά δεν βρίσκονται στο πλαίσιο ενός τέτοιου είδους κανονισμού. Ευχαριστώ. Thank you very much, um, έχετε ερωτήσεις προς τον ε, ομιλητή. Κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ καυτό το θέμα γιατί νομίζω το καλύτερο θα ήταν να διαγράφονταν αυτές οι παράγραφοι διότι αυτά που περιλαμβάνουν δεν φέρνουν τίποτα. Αν δεν είναι ρεαλιστικό πώς θα έχουμε αυτή την ε, συμμετοχή των ε, πολιτών ή ε, πώς θα ενδιαφέρονται οι διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων, ενδιαφερόντων αν δεν έχουν τη χρηματοδότηση. Πράγματι είναι καυτό το θέμα. Έχουμε το πρωτοβουλίες, όπως οι πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων Πολιτών που δείχνουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη μία αντιμετώπιση των διαστάσεων και των πτυχών όλων των παραγράφων. Εγώ δεν θα έλεγα να διαγραφούν η συγκεκριμένη παράγραφος τουλάχιστον, αλλά αν μείνει και πρέπει ε, συνειδητά να είναι ασαφής και εκτός κανονισμού να αντιμετωπιστούν με άλλους τρόπους σε σημαντικέ προκλήσει για να έχουμε μια συμμετοχή των πολιτών με νόημα. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να γίνει μια αναδιατύπωση. Ο στόχος μου βέβαια δεν είναι να διαγραφεί η πάνω επειδή είναι αυτό το θέμα, απλά να το χειριστούμε πιο επιδέξια και ίσως ε, σε διαφορετικό πλαίσιο. Πρόεδρος. Κάποιος άλλος. Πώς θα αποκτήσει νόημα δηλαδή είναι το θέμα. Εντάξει, πώς το παρόν το αφήνουμε εδώ. Όποιος έχει καλή ιδέα θα πάρει βραβείο, λέει κυρία Γκρέσλε. Προχωράμε. Έχουμε το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων από την Τσεχία ο πρόεδρος της μη κυβερνητική οργάνωσης από την χώρα αυτή που ονομάζεται Καλή Διακυβέρνηση ο κ. Λούκας Βάνιεκμερ. Έχετε το λόγο. Στα τσεχικά. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα να κάνω αυτή την παρουσίαση. Για μας είναι ένα άκρος επικαιρό θέμα, στι τελευταίες ημέρες. Ε, και ε, έχουμε πραγματικά έντονες αντιπαρθέσεις και ανταλλαγές απόψεων για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή μας για το νέο ε, κανόνα, αυτό θα είναι το πρώτο σημείο και έπειτα θα σας πούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα της σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Και μετά θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να δούμε πού είναι καλή αυτή η πρωτοβουλία και πού χρήζει βελτιώσεων. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων, αν δεν ξέρουμε ποιος παίρνει τις επιδοτήσεις ή τη χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα ερώτημα που με απασχολεί. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και συγκεκριμενοποίησης. Αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή η χρηματοδότηση, η ενίσχυση να πάει σε χέρια άλλα από αυτά στα οποία θα έπρεπε να πάει. Έχουμε και τα άρθρα 59-60 και θέλω να πω κάποια πράγματα που είναι σημαντικά. Ε, θετικό είναι που έχουμε τον ορισμό της οίκου συμφερόντων. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τους ε, υπαλλήλου. Πώς μπορούμε καλύτερα να αναγνωρίζουμε τέτοια ε, φαινόμενα, τέτοια κρούσματα. Επίσης υπάρχει, ε, είναι συστηματικό το ζήτημα, διότι πρέπει να δούμε ποιος είναι και ο τελικός δικαιούχος. Αν δεν ξέρουμε ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, δεν ξέρουμε αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή όχι. Γίνεται μια προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα σε επίπεδο αποδεκτών, δικαιούχων. Τι γίνεται με αυτούς όμως που είναι στα δημόσια μητρώα, αναφέρεται και το όνομά του είναι στα διάφορα συμβούλια. Ποιο είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης που ασκεί την επιρροή. Μόνο αν το γνωρίζουμε αυτό μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα. Γιατί πολλές φορές δεν είναι τα φυσικά πρόσωπα αυτά που αναφέρονται, τα πραγματικά, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και με αυτή τη ρύθμιση δεν το αντιμετωπίζουμε. να προσέχει και κάτι ακόμα. Το παιδί εφαρμογή κανονισμού για την σύγκρουση ε, συμφερόντων σε ό,τι αφορά του δημόσιου υπαλλήλου. Νομίζω ότι καλή περιγραφή γίνεται, αλλά σε ό,τι αφορά την ε, χρηστή διακυβέρνηση, θέλουμε να δούμε τι γίνεται στην πράξη. Και τι πρέπει να δημοσιοποιείται. Έγινε στο τέλος του χρόνου μια μελέτη με επτά επιχειρησιακά προγράμματα, περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Κάναμε την αξιολόγηση, είδαμε τις δομές ιδιοκτησίας και πραγματικά είναι σχετικά τα στοιχεία. 27% των χρηματοδοτηθέντων έργων είχαν ασαφή ιδιοκτήτη ή ε, μη κατονομαζόμενο το 38% σηματοδότηση δόθηκε σε έργα όπου ο τελικό δικαιός ήταν αφανή, ασαφή. Ε, δεν ήταν ξεκάθαρο Ποιο ήταν. Εμείς ε, στείλαμε και ερώτηση στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Budget και η απάντηση μας εξέπληξε. Έχω τα επιχειρήματα εδώ μπροστά μου. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Budget, από ό,τι μάθαμε, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να αναζητηθεί η δομή διοκτησίας. Και στην Τσεχία δεν είναι εύκολο γιατί έχουμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία για τις ε, νομιστέριες, αλλά το θέμα είναι αν η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ προπολογισμή έχει τη σχετική αρμοδιότητα, τι κάνει για την πράξη, ποια είναι τα συμπεράσματα που καταθέσαμε. τα αναφέρουμε στην έκθεσή μας, ε, στην επιστολή μας μάλλον, ε, στην ε, γάμα δέλτα Έχουμε ένα πρόβλημα. Πιθανή χρηματοδότηση τρομοκρατών ή οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι πραγματικός κίνδυνος. Συγκαλυμμένη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και άλλοι παράγοντες. Η χρηματοδότηση τώρα των ΜΜΕ είναι δυνατή αλλά κάποιες φορές ε, μέσα σε αυτή τη δομή μπαίνουν και κάποιες μεγάλες εταιρείες που δεν είναι πολύ εμφανείς η ε, συμμετοχή. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Προχωρώ στο εθνικό επίπεδο. Για την Τσεχία σας είπα ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ένα νέο νομοθέτημα, έχουμε ένα νέο νόμο. Έχει γίνει πιο αυστήρη λοιπόν η νομοθεσία. και στο πολιτικό επίπεδο με τους Έχουμε με τους αξιωματούχους. Υπάρχει και ένα πρόβλημα με τον ασαφή ορισμό των καταπιστευματικών ταμείων. Όταν ιδρύεται ένα καταπίστευμα στην Τσεχία, λόγω του νομικού πλαισίου που ισχύει, θα μπορούσε άμεσα ή έμεσα να επηρεαστεί η διοκτησία λόγω της, ε, του ορισμού, του πώς γίνεται ο ορισμός ε, των ε, μελών των ΔΣ. Δεν είναι αποτελεσματικό. Πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τώρα της προσπάθειας επίλυσης της 20 συμφερόντων. Θα σας δώσω παραδείγματα των τελευταίων πέντε ημερών. Είχαμε ένα πρόβλημα με έναν μικρό αποδέκτη. Το πρόβλημα ήταν οι προϋποθέσεις ε, για την, ανα... για τη χρηματοδότηση ενός έργου για την ισότητα. Η γυναίκα του συγκεκριμένου αυτού έκανε πολλά αιτήματα και το πρόβλημα ήταν ότι ο συγκεκριμένος κύριος είχε πρόσβαση σε πληροφορίες που είχαν να κάνουν ε, με τον ορισμό και τελικά αυτό συνιστά βέβαια σύγκρουση συμφέροντων. Ανακαλύφθηκε βέβαια αυτό το κρούσμα και ανελήφθη δράση, δηλαδή τα πράγματα εδώ λειτουργήσαν καλά. Αυτό πάντως βγήκε και στον τύπο και στα μέσα ενημέρωσης. Το δεύτερο θέμα ήταν ε, μια γεωργική επιδότηση. Ήταν ένας ε, διευθυντής, ένας μάνατζερ, Ε, σε έναν όμιλο ε, γεωργικών χημικών προϊόντων. Και δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρη η δράση τους ό,τι αφορά και τη χρηματοδότηση. Εγώ, από ό,τι ξέρω, ανακάλυψα ότι πήγε συμφερόντων ε, με το συγκεκριμένο. Και διορθώθηκαν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για διόρθωση 2%, καταλυσμό 2% των, των μέσων. Εμείς θέλουμε να υπάρξει επανόρθωση δεν πρέπει να είναι 2% η διόρθωση, 100% ήταν στην Τσεχία. Δεν λέω αν το 2% είναι καλό ή κακό. Θα πρέπει όμως οι κανόνες που εφαρμόζονται στις συμφερόντων να είναι ενιαίοι. Αλλιώς δεν θα έχει εμπιστοσύνη ο Τσέχος πολίτης όταν ε, είναι μικρές οι διορθώσεις ε, σε έργα που συμμετέχουν μεγάλοι όμιλοι και μεγάλη διόρθωση όταν συμμετέχουν μικροί ε, σκλήμακας δικαιούχοι. Πολλά λοιπόν έχουν ακουστεί και ένας υπουργό το 2008 είχε πάρει κάποια επιδότηση για ένα θέρετρο κέντρο ευεξίας. Και τέλος πάντων βγήκαν νέες πληροφορίες ε, χθες. Υπήρξε χειραγώγηση της πληροφόρησης ε, σε ό,τι αφορά το αίτημα κτλ. Δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτό ήταν απάτη ή δεν ήταν απάτη. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της έρευνας. Απλά θέλω να πω ότι καλό θα ήταν να υπάρχει έλεγχος όταν μάλλον υπάρχει έλεγχος των εν λόγω έργων, να είναι σαφές και ποιος κάνει τον έλεγχο. Από το Υπουργείο Οικονομικών που έκανε τον έλεγχο, στην προκειμένη περίπτωση, δυστυχώς ε, δημοσιοποίησαν ε, μια αίθουσα που έλεγε ότι δεν έγινε τίποτε λάθος. Δεν βρήκαν κάποιο σφάλμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει ανάλυση κινδύνων. Και τον έλεγχο πρέπει να τον αναλάβει η Κομισιόν στη συνέχεια. Το πρόβλημα, γιατί αυτό που δεν μας ενδιαφέρει είναι αντικειμενικός έλεγχος. Ο Υπουργός Οικονομικών εδώ ήταν και επικεφαλής ε, του οργάνου του ελεγκτικού. Και αποδέκτης και υπουργός. Ε, αυτά είχα να πω και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ερωτήσεις σας. Έχω μια ερώτηση για το θέμα που αναφέρατε ότι δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που είναι οι πραγματικοί αποδέκτες ε, των ε, χρηματοδοτήσεων, των επιδοτήσεων. Πραγματικά με εκπλήσει αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον τομέα της ε, καταπολέμησης ξεπλήματος χρήματος. Λέει ξεκάθαρα ότι σε όλους τους τομείς οι πραγματικοί δικαιούχοι ακόμη και αν ε, βρίσκονται στο, σε δεύτερο επίπεδο, αν είναι πίσω από 200 εταιρείε, ε, θα πρέπει να κατονομάζονται. Και μου κάνει εντύπωση που δίνονται χρήματα, χωρίς να είναι γνωστοί οι πραγματικοί δικαιούχοι. Αυτό με εντυπωσιάζει. Θεωρώ ότι Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να μην γνωρίζουμε σε ποιον έχουν δοθεί τα χρήματα. Και βέβαια έχουμε τα προβλήματα της χρηματοδότησης, τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος. Πώς θα τα λύσουμε αν δεν γνωρίζουμε τον ε, πραγματικό αποδέκτη, πώς θα καταπολεμήσουμε τέτοια κρούσματα. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Κυρία Κρέσλη, να προσθέσω και εγώ κάτι. Υπάρχουν κάποια μοντέλα ε, όπου έχουμε κάποιους ανώνυμους μετόχους σε κάποιες εταιρείες ε, και το έχουμε αναφέρει, το ρόλο αυτών των ανώνυμων μετόχων και είπαμε ότι υπάρχει και ένα ολόκληρο δίκτυο ε, διαφόρων κανόνων που λένε τι πρέπει να γίνεται και τι δεν πρέπει να γίνεται. Το πρόβλημά μας όμως ποιο είναι. Όταν έχουμε τέτοιες μορφές εθνικών εταιριών που προβλέπουν, ας πούμε, την και τα κτλ. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και στρέφομαι και στο ελεγκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά το ισοδύναμο πλήρων ελέγχων για τους οργανισμούς. Πρόεδρος, σας προτείνω εδώ και τώρα να ακούσουμε την απάντηση ή δυνατόν για αυτό το ερώτημα και μετά θα βρεθεί η επόμενη ερώτηση. Κύριος Λαζάρου. Ναι, δικαταφατικά. Α, βλέπω τα πρώτα να βάλουν στο τροπή. Κύριε Μάγερ. Κυρία Γιάλα, Γιάλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με σύγκρουση των συμφερόντων, ο κύριος Χολμάγερ θα μπορούσε να σας πει πολλές ιστορίες για κάποιου ε, επίτροπου. Ε, Απίστευτε. Τέλος πάντων, για τη σύγκρουση συμφερόντων σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες για το διάστημα, τις αερομεταφορές κλπ. Οπότε οι ίδιοι φορείς, η Επιτροπή για αυτά τα σχέδια και προγράμματα έχουμε κάποιους επαγγελματίε τόσο εξειδικευμένους που γίνονται σε τέτοιο επίπεδο εξειδίκευση, ούτε στα πανεπιστήμια δεν υπάρχουν. Και μπορούν να δουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα επιστοποίηση, ασφάλεια για ένα αεροπλάνο, α πούμε. Ε, και έτσι γίνεται στι αερομεταφορέ, α πούμε. Είναι κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Οπότε και εν προκειμένου υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη φάση που έχουμε ένα cooling των προτέρων, ένα cooling εκ των υστέρων, ούτως ώστε να πιστοποιηθεί η ασφάλεια των αεροπλάνων, η διαλειτουργικότητα για τους οδρόμους, ας πούμε. Και να είναι δυνατόν αυτό να αιτιολογηθεί όσο γίνεται με μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Και έτσι να μπορούν να βοηθήσουν σε αυτές τις υπηρεσίες αυτοί οι επιστήμονες, οι επαγγελματίες και να έχουν και αξιοπιστία. Για να μην υπάρχει πρόβλημα αφενός σύγκρουσης σε συμφερόντα και από να έχουμε τους πιο αποτελεσματικούς τέτοιους ειδικού για το αεροπλάνο, την ασφαλειά του, για κάποια άλλο μηχάνημα τέλο πάντων που θέλουν διαλειτουργικότητα. Γιατί πολλέ φορέ μιλάμε για σύγκρουση συμφερόντων, μιλάμε πάντα για κάποιο είδου ε, απαταιώνα. Και με τα κριτήρια όλα τα οποία επιβάλλουμε, εμποδίζουμε, βάζουμε ένα φραγμό. Αλλά όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους καλύτερους για αυτούς τους κλάδους που τους χρειαζόμαστε. Να μην έχουν αφενός σύγκρουση συμφερόντων και από την άλλη να που δουλεύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια που δουλεύουν για τα κράτη τους χωρί πρόβλημα. Ένα αυτό. Άλλο τώρα. Πώ αντιμετωπίζονται οι πολίτες σε αυτή τη λειτουργία αυτών των καταπιστευμάτων, ιδρυμάτων, τέλος των ταμείων. Οι επιλέξιμοι, οι ωφελούμενοι, αυτό το οποίο μας είπατε να μην πέφτουμε την παγίδα και δεν μπορούμε τελικά να κάνουμε τη διαχείριση. Και αυτό, το, το, το, αυτό, η ωφέλεια τελικά αυτών, είτε πρόκειται για απασχόληση ή για υποδομές ή για νοσοκομεία ή για ΜΜΕ, να μην υπάρχει η αίσθηση της ανισότητας ότι ο Γιώργος σε αλφα χώρα να παίρνει ό,τι παίρνει ένα γεωργός σε μια άλλη χώρα. Άρα έχουμε μπροστά μας δουλειά. Αυτό θα πρέπει να βρούμε. Και η ωφέλεια από αυτά τα ταμεία να είναι ε, να ανακατενέμονται όσο γίνεται με μεγαλύτερη ισότητα. Να μην δημιουργείται εντύπωση αδικίας για προθεσμικά όργανα και για την ωφέλεια εξ αυτού. Σας ευχαριστούμε για όσα λέει ο πρόεδρο, κύριε Βάνιγκνεχτ. Αυτά τα οποία μας είπατε αφορούν τις πιθανότητε ε, διαφθοράς και δεν μπορούμε να έχουμε ως αφετηρία την κατάσταση κατά την οποία αποκλείουμε 100% το να υπάρξει διαφθορά. Όμως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε τουλάχιστον να έχουμε στεγανή ρυθμίση όσο γίνεται. Σύμφωνα το πρόγραμμα θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τις ερωταπαντήσεις και τη συζήτηση εδώ και 10 λεπτά. Αλλά μια που ήταν τόσο αξιόλογη η συζήτηση τόση ώρα, σας προτείνω το εξής από όλα αυτά τα αυτά θέματα που μας έμεινε ο κ. Βάγκεγνεχτ να πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, αλλά πρέπει να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βάγκεγνεχτ, λέει η κυρία Γκρέσλε. Αλλά θα πρέπει και το Συμβούλιο να μας ε, πει την άποψή του μια που εμπλέκεται σε όλα αυτά. Οπότε πιέζει ο χρόνος. Άρα, προτείνω να αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επιτροπή και όταν ο κύριο Βατίνη να δευτερολογήσει και εγώ θα ήθελα κάποιε απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Πώ είναι δυνατόν, δυνατόν όλα αυτά να ε, ισχύουν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ελπίζω ότι επίση θα υπάρξει ο χρόνο να μπορέσω να απαντήσω σε κάποια από αυτά τα οποία ακούσαμε από του προηγούμενου. Τώρα για αυτό το τελευταίο που είπατε για την ε, ε, σύγκρουση συμφέροντα και εγκληματική δραστηριότητα, αυτό το οποίο αναφέρθηκε πολύ σημαντικό, ξέλυμα χρήματο, είναι διαφθορά. Τι είναι, τι, άλλο, τι, τι είδου εγκληματικότητα είναι αυτή, υπάρχουν ε, κάποιοι ξεκάθαροι κανόνε και είναι ξεκάθαρε οι απαγορεύσει για τον ιδιωτικό τομέα σε τέτοιες περιπτώσεις να λαμβάνει η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε το άρθρο 106 του Οικονομικού Κανονισμού για το τι γίνεται με τους ε, ε, επιλέξιμους και υπάρχουν επίσης διατάξεις για το πώς η Όλαφ μπορεί να δει ε, ποιος κρύβεται πίσω από κάθε χρηματοδότηση να δούμε αν υπάρχει δραστηριότητα για να υπάρχει έλεγχος επ' αυτής της ε, εταιρείας. Οπότε υπάρχουν, ναι, κανόνες, υπάρχουν νόμοι για να υπάρχει πρόληψη των ε, εγκλημάτων αλλά και καταστολή τους. Και αυτό γίνεται με κώδικα διοντολογίας όσον αφορά κάποιες ε, υπηρεσίες ή γίνεται με την εθνική νομοθεσία. Επομένως, υπάρχει πρόληψη αλλά και από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει δημοτική δραστηριότητα η όλα αυτά ε, ασκεί κάποια έρευνα και μπορεί κάποιος να αποκλειστεί επί μία τριετία από τη χρηματοδότηση. Αλλά βέβαια συντρέχουν επίσης και οι ποινικέ διατάξεις του εθνικού δικαίου. Για τα άλλα θέματα τώρα. Να σας τα πω τώρα ή θέλετε να επανέλθω μετά. Συνεχίστε, συνεχίστε. Επ' αυτόν που είπε το ελληνικό συνέδριο σας τονίζω ότι θέλουμε να έχουμε σύστημα αναφορών πρώτα πρώτα για το σχέδιο προπολογισμού αλλά και για την απαλλαγή. Χρειάζεται εκεί. Δεν θα πρέπει να έχουμε επικαλύψεις, οπότε θέλουμε να υπάρχει κάποιο είδους δέσμη ε, εκθέσεων και έτσι να λαμβάνεται σχετική ενημέρωση. Τώρα όσον αφορά επιδόσεις, απόδοση, μεγάλη ιστορία, συμμετοχή των κρατών μελών, συνένεση μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων θεσμικών οργάνων. τι σημαίνει αποτέλεσμα, τι σημαίνει σχετικά με, το, με τα προσδοκόμενα, τα deliverables, παρακολούθηση της πρόοδου και αναφορά των όσων επιτέχθησαν. Έχουμε επίσης ε, αποθεματικό απόδοσης και έχουμε επίσης και καταβολές επί τη βάση αυτών των επιδόσεων. Νομίζω ότι πρόκειται για θέματα στο οποία πρέπει να είστε ενημερωμένοι. Να μπορείτε να λάβετε εσείς πολιτική απόφαση και να μείνει το σύστημα αυτόματο. Να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα και τις ενισχύσεις και το σύστημα παρεμβάσεων. Ο σκοπό είναι το πώς θα απλουστευτεί, θα διευκολυνθεί ο συνδυασμός των διαφορετικών μέσων στις σχετικές περιπτώσεις. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφές ότι αυτή η πρόσφατη κρίση απέδειξε ότι χρειάζεται ευελιξία. πόσο διάφορες, ε, διάφορες προτάσεις και είπαμε για τη μαξιλάρι πρέπει να υπάρχει, τι πρέπει να κάνουμε με τα καταπιστεύματα κλπ. Δεν είναι το θέμα ποσότητας χρημάτων, αλλά το τι θα κάνουμε με τα χρήματα που έχουν διατεθεί επί τη βάση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρέπει να είμαστε όσο είναι πιο αποτελεσματικοί. Αν χρησιμοποιήσουμε τα καταπιστέματα, Όπω ορθώς αναφέρθηκε, είναι γιατί στον προπολογισμό δεν προβλέπεται κάποια δαπάνη. Μπορεί κανεί να πει βέβαια ότι εμείς δεν χρησιμοποιηθήκαμε σωστά τα καταπιστεύματα. Υπάρχουν για τη Γεωργία Αφρική, για τη Λιβύη, για διάφορες περιοχές της χώρας. Για να κάνουμε κάτι για τις αιτίε της μετανάστευσης. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρησιμοποιήσει ορθά τα καταπιστεύματα. Έχουμε πει ότι πρέπει να αυξηθούν οι αρμοδιότητες της αρχής του προϋπολογισμού τώρα όσον αφορά τον ε, κανονισμό. Είπαμε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα νομοθετήσουμε για την μετά το 2020 περίοδο. Τα είπε ο Και οι εισηγητές ότι χρειάζονται κοινέ διατάξεις. Όσο γίνονται καλύτερες σε αυτόν τον κανονισμό. και σε αυτή τη φάση δεν μπορεί παρά να έχουμε κάτι σαν εργαλειοθήκη. Θα έπεται το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα το συζητήσουμε στην ώρα του. Κατόπιν η εμπλοκή των πολιτών. Σωστά ελέγχθη ότι υπάρχουν κάποια υπέρ για την εμπλοκή των πολιτών και άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε, το θέλουμε κάτι θετικό, να είναι κατανοητό. Τόσο αφορά την κατανομή των πόρων, θα πρέπει να δούμε την ευκαιρία να είναι πιο αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απλούστευση να μην είναι πρόφαση και οι υπηρεσίες θα πρέπει να υποστούν τέτοιου είδου κατανομή να συνεργαστούμε για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να έχουμε και εξοικονομήσεις δαπανών. Δεν ξέρω πω θέλει ο συνάδελφο να συμπληρώσει τα όσα σας είπα. Ή συνάδελφος. Αυτά τα ταμεία τα οποία ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι, όπως είπε και η Ολίβια, ο στόχος για το 2014-2020 στην νομοθεσία ήταν να δώσουμε μια σειρά από εναλλακτικέ λύσεις, εργαλεία για τις διαχειριστικές αρχές να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν ένα είδος βοήθειας, επιδότηση, επιχορήγησης, ε, δανείου που αποπληρώνεται κτλ. Και όλα αυτά να δίνονται ως εναλλακτική λύση και το νομικό πλαίσιο να είναι πάρα πολύ πλήρες και σαφές. Δεδομένη των δεδομένων των επικρίσεων που ακούστηκαν, που είπαν ότι λείπουν στοιχεία και οδήγησαν στα προβλήματα τα οποία ακούσαμε ακόμα και σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της τροποποίησης αυτής προσπάθησε στα πλαίσια της ενδιάμεσης αξιολόγησης, γιατί εκεί βρισκόμαστε και όχι στο μετά το 2020, να βελτιώσουμε την κατάσταση με στοχευμένο τρόπο, χωρίς όμως να ανατρέπουμε πλήρως την κατάσταση και να δώσουμε και επιπλέον ε, εναλλακτικέ λύσεις ε, στις διαχειριστικές αρχές και ένα συνδυασμό είναι το FCSIF. Και έτσι θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε και το ΕΦΣΙ σε κάποιες περιοχές των κρατών μελών όπου η εφαρμογή δεν ήταν τόσο υψηλή σήμερα. Στα πλαίσια αυτή τη διαδικασία ακούσαμε μια ιδιαίτερη προσοχή στις διαχειριστικές αρχές που εφαρμόζουν εδώ και κάποιο χρόνο αλλά όπως επίσης και στην, υψηλή, στο, στην ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλούστευση και στο το τομιακό κομμάτι των αλλαγών θα δείτε πως έχουμε μια σειρά από ενημερωμένες αναφορές στον κανονισμό και εδώ έχουμε συμπεριλάβει και τη σύγκρουση συμφερόντων για παράδειγμα. Ευθυγραμμιζόμαστε λοιπόν με τη γενικότερη προσέγγιση να προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συνεκτικοί και συνεπείς στις προσπάθειες που κάνουμε. Ωραία λοιπόν. Αυτή ήταν η σύνοψη Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Σας παρακαλώ πολύ δείξτε υπομονή στον τρόπο που σκέφτομαι. Πριν δώσω το λόγο τώρα στους δύο συγητές για τα προσωρινά συμπεράσματα, θα ήθελα να επιστρέψουμε σε ένα προηγούμενο ομιλητή, γιατί σε 15 λεπτά θα φύγουμε από την αίθουσα και θα αναρωτιόμαστε πώς, όταν πια θα υπάρχουν ε, ε κανόνες, αν αυτοί οι κανόνες θα είναι πραγματικά ισχυροί ή όχι ή θα μπορεί κανείς να τους παρακάμψει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε διάφορα. Πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν να γίνουν πιο αυστηροί και σε πρακτικό επίπεδο οι κανόνες αυτοί ή τι. Já bych určitě nerozporoval, že Evropská komise pravidla nastavená má, nicméně podle mého názoru nejsou dostatečně implementována jak na evropské, tak i národní úrovni έχει καθορίσει κανόνε. Θα ήθελα να σα πω πω σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, αλλά θα πρέπει να το δούμε και σε ευρωπαϊκό, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Δεν έχουμε την πλήρη μελέτη. Έχουμε εδώ δικαιούχου οι οποίοι δεν επαληθεύθηκαν και δεν αξιολογήθηκαν καθόλου αυτή τη ε, διαδικασία. Έχουμε πληροφορίε που μα οδηγούν στο εξή συμπέρασμα. Για μια φορά ακόμα πρέπει να γίνουν επαληθεύσει γιατί οι επαληθεύσεις αυτές βασίζονται στις δηλώσεις που έχουν υποβάλει μη συμφερόντων. Και ε, εγώ πρέπει να σας πω πως κατέθεσα τα έγγραφα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας είπε πως δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Εάν υπήρχε μία μέθοδο συγκεκριμένη για να γίνει αυτή η επαλήθευση, θα μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτές τις δηλώσεις. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να δούμε τι προτείνουν και τα κράτη. Να σας πω πως στην δημοκρατία της Τσεχίας το θέμα της χρήσης και της κατάχρησης των διασωτικών ταμείων είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ευρύτερα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για την ε, τσεχική δημοκρατία ναι, ισχύει αυτό που σας λέω. Επίσης, η προθεσμία που θα ε, διδετε, δηλαδή μέχρι να θεωρήσουμε πως υπάρχει, ε, υπάρχει ένδειξη απάτης ένα χρόνο, δύο χρόνια, ε, νομίζω ε, σε αυτό το διάστημα το κράτος μέλος που αναμένει να του χορηγηθούν κάποια κονδύλια δεν θα πρέπει να τα λαμβάνει και θα πρέπει να δει όχι μόνο την αυτοδιαχείριση, την ίδια διαχείριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά να δει τι κάνει και κάθε μεμονωμένο έργο γιατί θα πρέπει να δούμε μέχρι ποιο βαθμό, μέχρι ποιο βαθμό έχουμε σύγκρουση συμφορώντων η οποία ενδεχομένως θα έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις και τότε ήθελα να στραφώ προς το Συμβούλιο. Ναι, το είπα και εγώ. Οπότε, σας παρακαλώ πολύ, κάνα δύο λεπτά τη δική σας άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους. Θα ήθελα καταρχήν να σας συστηθώ. Λέγομαι Γκίλτ Φλόρες και είμαι αυτή τη στιγμή στην Προεδρία της ομάδας στο Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή Είμαστε στην κατάστρο εξέταση του, της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή τη στιγμή κλείνει η πρώτη εξέταση. Πού θα ακολουθηθεί από προτάσεις για οποιαδήποτε αλλαγή προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινήσαμε αρχές Ιανουαρίου. Ε, κοιτάμε όλα τα άρθρα ένα-ένα. Άρα λοιπόν Ελπίζουμε πως θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τα τέλη της Προεδρίας μας. Έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή για, το, για τον τρέχοντα κανονισμό, οικονομικό κανονισμό, τον οποίο ε, περιμένουμε ε, να εξετάσουμε για να παρουσιάσουμε μετά τις συμβιβαστικές μας τροπολογίες του επόμενους μήνες. Με χαρά θα συνεργαστούμε μαζί σας, μια και είστε ο έτερος διαπραγματευτείς. Αυτά. Ναι, να μια σπάνια ευκαιρία να σας κάνουμε λοιπόν ερωτήσεις εδώ. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Πότε θα έχουμε μια ε, συνολική θέση, πιστεύετε, από πλευράς ε, Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή συντονίζουμε τις εργασίες και διατυπώνουμε το πρώτο, το πρώτο τμήμα για τα πρώτα άρθρα των συμβαστικών κειμένων. Να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει αυτό στο ίδιο το Συμβούλιο και μετά θα το δείτε και εσείς με λεπτομέρειες. Οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τον οδικό χάρτη που έχουμε θέσει τον Νοέμβριο και για τον οποίο είμαστε ακόμα σε επαφή και, που μας και με τον οποίο μας βοηθήσατε στην αρχή της Προεδρίας. Ναι. Θέλουμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε τις προθεσμίες του οδικού χάρτη. Ελπίζουμε λοιπόν πως μπορεί να έχουμε κάποια καθυστέρηση. Ότι ακόμα και αν έχουμε κάποια καθυστέρηση θα σας στηρίσουμε ενήμερες, αλλά ελπίζω πως όχι. Excellent. Any other questions? Okay. Άλλες ερωτήσεις. Ωραία. Στην αρχή της συνάντησης ξεκινήσαμε με την κυρία Γκρέσλερ. Έπια, για να είμαστε δίκαιοι, να ξεκινήσω με τον κύριο Άσχουτ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί πιέζει ο χρόνο. Αλλά σα υπενθυμίζω ευθύ εξ αρχή ότι ο στόχο όλων αυτών ήταν το πώ θα μειώσουμε τη γραφειοκρατία, για την πολυνομία, πώς θα έχουμε καλύτερα ποσοστά σφάλματος στον προπολογισμό και επίσης όσον αφορά το ότι ε, υπάρχει σχέση μεταξύ πολυπλοκότητας και ποσοστού σφάλματος, ε, γι' αυτό θα πρέπει να ενεργήσουμε. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι το πώς θα βελτιωθεί η πρόσβαση στον προπολογισμό την ώρα των αποτελεσμάτων και την ώρα που έρχεται η στιγμή να καλυφθεί ο πολίτης. Ελέγχθησαν κάποια πάρα πολύ σημαντικά, ιδίω όσον αφορά το πόσο θα πρέπει να στεγνώ το σύστημα, ιδίω όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, πολύ ενδιαφέροντα και ε, επίση και την εμπλοκή των πολιτών σχετικά με τον προπολογισμό, όπω προηγουμένω τα συζητήσαμε. Αυτό πάντοτε με έχει προβληματίσει. Έχουμε εκατοντάδε εκατομμυρίων που θα πρέπει να μην αισθάνονται μακριά. Γιατί είναι πενταετή η θητεία. Είναι το θέμα της υποχρέωση λογοδοσία επίση με τον προπολογισμό. Και εκεί πάντοτε υπάρχει πρόβλημα. Άρα θα πρέπει αυτό να το δει το κοινοβούλιο, να το επιλύσει. Είναι περίπλοκη αυτή η δουλειά μας και αυτό το είπανε πολλοί ομιλητές. Οπότε ειλικρινές ευχαριστίες σε όσους ήρθαν, το υλικό που μας έδωσαν, που μας μίλησαν, ήταν όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστίες και προς τους συναδέλφους και όσους έχουν απομείνει στην αίθουσα. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις τους και θα προσπαθήσω να καλύψω τα όσα σχολίασαν. Έχεις το λόγο, Ίγκα. Έχουμε κάποια λεπτά ακόμα. Έχουμε αναφέρει πλέον και σε επιτάπητος και ορισμένα άλλα προβλήματα που τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μάλλον θα κατατεθούν και άλλες τροπολογίες. Αλλά πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω ε, όλους που είστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και το θεματικό τμήμα ε, την ε, γραμματεία της Επιτροπής μας και της ε, Επιτροπής προπολογισμών. Ξέρω επίσης και ότι οι συνεργάτες μας είναι και αυτοί πολύ άσχολοι. Νομίζω ότι καλό θα ήταν η Κομισιόν να μας δώσει κάποιες παραπάνω πληροφορίες σε ό,τι αφορά πέρα τον κανόνα για τη μία αποκόμιση κέρδους η συνολική κατάργηση ίσως να μην είναι λύση ή θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση. Να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ μικρών μεγάλων, ομίλων, ε, μη κερδοσκοπικών και κερδοσκοπικών Καλό θα ήταν να γίνει μια καλύτερη διαφοροποίηση, δηλαδή ναι να υπάρχει απλούστευση, ε, αλλά να μην δώσουν προς τα έξω την ε, εικόνα ότι ε, επιτρέπεται η αποκόμιση κέρδους με χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Νομίζω αν μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση θα είμαστε ήδη στο σωστό δρόμο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάποια τελικά σχόλια. Είναι αδύνατο να συνοψίσει κανείς καταρχήν τα όσα άκουσε. Ήταν πραγματικά τεράστιος ο κατάλογος. Και ίσως πιο προβληματικό γίνεται από το γεγονός ότι τα όσα συζητάμε δεν είναι συγκρίσιμα σε πολλές περιπτώσεις. Και δεν μπορούν να συγκριθούν ε, μεταξύ τους γιατί μιλάμε για διαφορετική διάσταση. Οπότε το κατά πόσο έχουμε τις αυτές τις μεγάλες, μεγαλεπίβολες ιδέες για την απλώς, απλούστευση, ε, για την ε, ε, μία ενιαία αναφορά, όπως είπε το Ελληνικό Συνέδριο, την κατάρτιση προϋπολογισμού βασίστες σε επιδόσεις, τους χρηματοδοτικούς κανονισμούς, μη κέρδος, εσωτερικά καταπιστεύματα, ευελιξία. Είναι όλα λοιπόν πολλά μαζί στην κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι τεράστιο το θέμα. Και μια τελική σκέψη. Και δυστυχώς θα συμφωνήσω με τον κύριο Νούνιες Φερέρ, παρόλο που δεν χρησιμοποιήσει αυτά τα λόγια. θα τα πω εγώ όμως τολμηρά και επιτρέπετε. Δημιουργήσαμε ένα τέρας. Πραγματικά δημιουργήσαμε ένα τέρας. Και η τεράστια πρόκληση μπροστά μας είναι εμείς πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και πρέπει πραγματικά ο λαός της Ευρώπης θα πρέπει να ενδιαφέρεται και να προσέχει και να σέβεται ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε. Αλλά εδώ χρειάζεται η συμμετοχή, η εμπλοκή των πολιτών. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τη σύγκρουση συμφερόντων, το παραδοσιακό κομμάτι που συζητάμε τόσα, τόσο καιρό, αλλά και την απλή σκέψη πως υπάρχει δυνατότητα πραγματικής απάτης χωρίς κανό, καν κάποιος να το καταλαβαίνει. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε φωναχτά. Αυτό θέλουν οι πολίτες της Ευρώπης. Αυτό τους ενδιαφέρει. Θα πρέπει να τα καλύψουμε λοιπόν όλα και όπως είπα Τυχερά δεν, είμαστε τυχεροί, δεν είμαστε μόνοι, είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει όλα αυτά να τα δρομολογήσουμε. Σας ευχαριστώ για μια τόσο καρποφόρα συνάντηση, σεμινάριο. Να συνεχίσουμε λοιπόν τις προσπάθειες και πριν φύγετε από την αίθουσα να σας υπενθυμίσω πως αν σας ενδιαφέρει και έχετε ακόμα κάποιες δυνάμεις, κατεβείτε δύο ρόφους στο 2Q2 στην αίθουσα αυτή θα έχουμε μία μεικτή συνάντηση με τις Επιτροπές ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιωσιμή Ανάπτυξη. Ένα ακόμα ταμείο που θέλουμε να στήσουμε. Ίσως. Ευχαριστώ.